Καταρχά, καλημέρα σα. Το διαπραγματευτικό, τη διαπραγματευτική εντολή για την έκθεση του κυρίου Φλέκενστάιν. Οι συντονιστέ, συμφώνησαν στο αίτημα του κυρίου Φλέκενστάιν να αρχίσουμε τι διαβουλεύσεις μαζί με τους, ηγητές και το, με τους και το Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση υιοθετήθηκε το Δεκέμβρη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ωραία. Ως πρόεδρος λοιπόν θα δώσω το λόγο στον... Μάλλον θα δώσω την εντολή στον κύριο Φλέκενστάιν για όλους αυτούς τους τομείς τους οποίους χειρίζεται και έχει την εντολή να κάνει τη διαβούλευση με τους κοιόδης ηγητές και το Συμβούλιο. Δεύτερον, ορισμός εισηγητών και συντακτών τρεις ε, εκθέσεις στο πακέτο της ε, αεροπορι... των αεροπλάνων. The introduction. Αεροπορικές σχετικά με τη μείωση των θορύβων σε, ε, αεροπλάνα, σε αεροδρόμιο της Ένωσης. Δεύτερον, κοινές, ε, κοινοί κανονισμοί για τα σλότς, πάλι σε EU ε, αεροδρόμια, ALDE και ανακύρωση της ε, οδηγίας 90-97 ΕΛΚ. Γνωμοδοτήσεις τώρα αποφατητήσαμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τις προτάσεις του Συμβουλίου που καθορίζει ε, το, την αύξηση μέχρι το 2020 σε μία γνωμοδότηση. Ενώσουμε τις δύο γνωμοδοτήσεις και αυτή θα πάει στο ALDE στο 6 μηχανισμοί για τα αέρια του θερμοκηπίου ε, σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Οι συντονιστές μας προτείνουν καμία δράση, ουδεμία δράση. Επίσης, στη συμφωνία μεταξύ EU και USA, ε, επειδή γίνεται από την ομάδα των ε, δομικών ελευθεριών, καμία δράση, αλληλεία και ταμείο αλληλείας καμία δράση για το σύστημα, το δορυφορικό, ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα αποφασίστηκε να κάνουμε μία γνωμοδότηση και αυτή θα πάει στην ECR, Ευρωπαϊκή Συντηρητική. Η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ουδεμία δράση, ουδεμία ενέργεια. Ε, για τα multi vehicles η απόφαση είναι να κάνουμε να δώσουμε μία απόφαση και αυτό θα το πάρει κυκλικά και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την πολιτική των αεροδρομίων η απόφαση ήταν καμία ενέργεια διότι όλο αυτό θα καλυφθεί από τις τρεις στο πακέτο, τις τρεις νομοδοτήσεις στο πακέτο δηλαδή. Επίσης το πρόγραμμα εργασίας 20 12 καμία δράση διότι ξέρουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας θα αποφασιστεί στην Ολομέλεια. Ανακοίνωση της Κομισιόν για την ανάπτυξη ναυτιλιακής στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού. Οι συντονιστές πιστεύουν ότι θα πρέπει να εκδώσουμε μία γνωμοδότηση σοσιαλιστές και δημοκράτες μετά η ετήσια αύξηση, ε, ανάπτυξη, ε, καμία, ουδεμία ενέργεια, όπως σας είπα, Κομισιόν 2020, αυτό συνδέεται με το Φόρουμ 5, ουδέμια δράση εδώ, ουδέμια ενέργεια, διότι καλύπτεται με τα προηγούμενα σημεία. Επίσης, ουδέμια ενέργεια στα, στα, δύο ανακοινώσεις, το άλλο το μελλοντικό ΦΠΑ και ε, εδραίωση ενός ε, δυνατού συστήματος ΦΠΑ και η κοινή απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ε, της, ε, το παράρτημα 13 EEA, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για το ECOL για ε, την ασφαλή διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης ε, υπό τις ε, διατάξεις της οδηγίας ITS. Επίσης πρότειναν να κάνουμε κάτι για το e αργότερα. The Επίσης, ο Πρόεδρος ανα, συζήτησε με τους συντονιστές το εξής ότι η Ουγγαρία θέλει να αλλάξει το ενεργειακό και λειτουργικό πρόγραμμα και οι συντονιστές αποφάσισαν να, να αρχίσουν διαβουλεύσεις διότι οι δύο συναρμόδιοι επίτροποι αντιτίθενται στο, στην πρόταση αυτή της Ουγγαρίας. Επίσης, Έχουμε μία επιστολή που υπογράφει από 24 ευρωβουλευτές που ε, αντιτίθεται στο οδικό ε, πρόγραμμα Λιόν Τουρίνου ε, και τα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην Ιταλία με τις αστυνομικές αρχές, τις διαδηλώσεις κλπ. Και συμφωνήσαμε να προτείνω να να στείλω μία επιστολή στον κύριο Μπρίνκχορστ και να ζητήσω λεπτομερείς πληροφορίες από εκείνον για το θέμα αυτό. Τι γίνεται με αυτόν ε, την πρόταση του, του, αυτοκινητόδρομου ή των μεταφορών τέλο πάντων μεταξύ Λιών του Ρήνου. Και όταν θα έχουμε αυτή την απάντηση οι συντονιστές θα κάνουν μία συζήτηση ε, εις βάθος ε, ε, σχετικά με την επιστολή αυτή των παραπώνων των 24 Ευρωβουλευτών. Θα συζητήσουμε λοιπόν στο πλαίσιο των συντονιστών αυτή την επιστολή αργότερα. Αυτά ως προς το περιεχόμενο των συντονιστών, εχθές, τη συζήτηση των συντονιστών. Ο κύριος Αλ Καντράουι. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Κράμερ να μας φωτίσει ο κύριος Κράμερ. Τότε οι δύο συντονιστές για τα TENS, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, είχαν συμφωνήσει εάν οι δύο μεγάλες ομάδες πάρουν τα δύο αυτά μεγάλα ντοσιέ να προτιμήσουμε συνεχεία τις άλλες πολιτικές ομάδες στο πακέτο των, ε, αεροπορήτων των αερομεταφορών. Και είχε εσύ τότε ότι οι μικρότερες εμάδες μπορούν να έχουν μια κατανομή των ε, εξαίσεων στο θέμα του, του αεροπορικού πακέτου. Ε, αυτό ήταν σαφές για τους φιλελεύθερους. Ε, συνεχεία όμως μας είπες ότι όχι, αυτό είναι λάθος. Ε, διότι οι συντονιστές πήραν μεν μία απόφαση, αλλά την ακύρωσαν αργότερα. Αυτό δεν το βρίσκω σωστό, δεν είναι δίκαιο και γι' αυτό ζητώ να πάρουμε εμείς τον ντοσιέ ξανά. Να τηρηθεί η παλιά υπόσχεση. Μάλιστα, τώρα δίνω το λόγο, λέει ο πρόεδρος, στον κύριο Αλκαντράουι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί μια μικρή σύγχυση εδώ. In ε, Πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι στην κατανομή των δύο εκθέσεων. και για την έκθεση για τη χρηματοδότηση. Κανονικά λοιπόν θα πρέπει να ορίσουμε δύο εισηγητές από τις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες Στη συνέχεια θελήσαμε να κάνουμε, θα έλεγα, μια καλή πράξη και είπαμε ας μη μονοπολούν κάποιοι τα πράγματα και ας δώσουμε τη δυνατότητα και στην επόμενη πολιτική ομάδα, η οποία είναι μικρότερη, ας της δώσουμε την τιμή λοιπόν να έχει μια κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα θέματα αυτά για, τα, για τους αερολιμένες. Εμείς ξεκινάμε από από την αρχή ότι οι φιλελεύθεροι θα μπορούσαν να κάνουν την επιλογή της και μετά οι άλλες δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες θα ε, έβλεπαν μεταξύ τους τι θα γίνει ε, με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, τις μικρότερες. Έχουμε περισσότερους πόντους από τους πρασίνους και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση. mijn voorstel zou zijn eh, αυτό το οποίο λοιπόν σας προτείνουμε μετά τη συνεδρίαση να συζητήσω με τον Μάικελ προσωπικά και αν υπάρχει πραγματικά λόγος να επανέλθω στη συζήτηση. Και να σας προτείνω λοιπόν Μάικελ μια συζήτηση μήπως ε, αλλάξει κάτι. Προς το παρόν όμως εμένω στην απόφαση η οποία λήφθηκε χτες. Oh, oh. Can I, before I bring you... Πριν... Πριν σας δώσω το λόγο, πρέπει να ξέρουμε Ποιο θα κάνει αυτή την έκθεση. Η πρόταση είναι να μείνει σοσιαλιστέ και δημοκράτες, αλλά κάνετε μια, κάντε μια κουβέντα γρήγορα, κουβεντιάστε το, ταχύτερα, ε, διότι εδώ προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ένα κοινοβούλιο. Ο κύριος Αλκαντρούη. Προτείνω να το κάνω αυτό σήμερα, να κάνω αυτή τη συζήτηση και στο, προς το τέλος της συνεδρίασης θα πληροφορήσω τη γραμματεία για την απόφαση. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Εμείς συζητάμε τα πράγματα μεταξύ μας και είμαστε, εγώ είμαι από μια μικρότερη ομάδα και θα ήθελα να δω περισσότερες ευκαιρίες για την ομάδα μου και θα ήθελα να έχω περισσότερες γνωμοδοτήσεις, περισσότερους εισηγητές. Όλοι μπορούμε τώρα να γκρινιάζουμε και να παραπονιόμαστε, <clears throat> αλλά το θέμα είναι ήρθε η σειρά μας και πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε, τι μπορούμε να λάβουμε ως εισηγητές, ως κοιόδης. Πιστεύω ότι η ομάδα μου είναι πολύ ευτυχής να διαβουλευθεί με το ε, ΕΛΚ, με τους συντηρητικούς, με την Άλντε, όταν έρθει η ώρα κατανομής των γνωμοδοτήσεων. Αλλά δεν ήξερα ότι αυτή είναι η διαδικασία την οποία εφαρμόζουμε. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, έτσι είπαν οι συντονιστές, έτσι συμφωνείς και τώρα αν αυτοί θέλουν να παραιτηθούν έχει καλός. Προς το παρόν όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα το ταχύτερο να ξέρω αν υπάρξει κάποια αλλαγή για να προχωρήσουμε. Προτείνω λοιπόν οι σοσιαλιστές οι δημοκράτες και οι πράσινοι να συζητήσουν. Ο κύριος Βαντάλεν. Μία συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Αλκαντράουι. Πράγματι θα πάρει το καφεδάκι του και θα συζητήσει το θέμα για τη συγκεκριμένη έκθεση. Αλλά γιατί θα πρέπει να το συζητήσει με τον κύριο Κράμερ και όχι μαζί μου σαν παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι θέλει να το δώσει στον κύριο Κράμερ, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι ακριβώς συμφωνία έγινε μεταξύ των συντονιστών. Εδώ έχουμε μία <clears throat> ασυμφωνία, δεν έχουμε σύμπτωση απόψεων. Και όπως είπε η κυρία Φώστερ πολύ σωστά, έχουμε ένα σύστημα το οποίο πάει ανάλογα με... We even, we have a system that some of the committees don't. Ανάλογα με πόντους. Όποιος πάρει, πάρει τους μεγαλύτερους πόντους παίρνει και την έκθεση. Τώρα έχουμε ένα σύστημα όπου μπορεί να έχεις μία μόνο επιλογή επιλογή. Ο κύριος Αλκαντράι εφάρμοσε ή μάλλον χρησιμοποίησε αυτή την ευκαιρία, αλλά έχει το δίκαιο να ανακαλέσει, να αλλάξει γνώμη. Δεν θέλουμε την έκθεση και την ξαναβάζουμε στην κοινή δεξαμενή των πόντων. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα γίνει αλλαγή ή όχι. Ο κύριος Κράμερ. Κοιτάξτε, εδώ δεν πρόκειται να κλείσουμε μια συμφωνία και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Συνήθως, κάθε έκθεση έχει έναν ραπορτέρ. Και στι μεγάλες εκθέσει είχαμε συμφωνήσει δύο εισηγητέ. Εντάξει. Είχαμε πει θα δώσουμε τις μεγάλες εκθέσεις, τις μεγάλες ομάδες, αλλά στον επόμενο γύρο θα δώσουμε εκθέσεις στις μικρές ομάδες. Αυτό ήταν το deal, αυτή ήταν η συμφωνία μας και ε, χτες τι έγινε και τι δεν έγινε μπορούμε να το, συζητήσουμε αλλά φαίνεται τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Ο πρόεδρος. Είναι έκθεση σοσιαλιστών και, και ε, δημοκρατών. Okay. Ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών. έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, η ομάδα, η σοσιαλιστική ομάδα έχει επίσης ακόμα ένα πόντο συν ένα, διότι ήταν 11 ενώ τώρα είναι 12 μετά την ολιμέλεια που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ε, άλλο πόντο προς όφελός τους. Μάλιστα, Επόμενο θέμα. Πριν αρχίσουμε με την ψηφοφορία, χρόνια πολλά στον κύριο Φλέκενστάιν. 31 Είναι ο, ένας μπέμπις 31 ετών. Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τελευταία μέρα που θα έχουμε την κυρία Κάσνιτς ως ε, επικεφαλής της γραμματείας. Η κυρία Κάσνιτς θα μας αφήσει στο τέλος του χρόνου, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία που εμείς όλοι τη βλέπουμε σε αυτή την εξέχουσα θέση που κάθεται εδώ μαζί μου. καμιά φορά κουνάει το κεφάλι της με τα απίστευτα που ακούει, άλλες φορές τα κουνάει, κουνάει το κεφάλι της συγκαταβατικά ή με ευχαρίστηση. Εν πάση περιπτώσει ήταν χρόνια στην Επιτροπή μας και της είμαστε λίγαν ευγνώμονες για την εργασία που έχει κάνει, η οποία ήταν εξαιρετικά επαγγελματική. Ε, έχοντας λοιπόν υπόψη αυτό το γεγονός, θα διανύμουμε ένα βιβλιαράκι το οποίο δεν είναι συλληπιτήριο προς Θεού, αλλά τα μέλη θα μπορέσουν να υπογράψουν στο βιβλίο αυτό ή να γράψουν ε, κάτι αναμνηστικό. Ε, και καταφέραμε να βρούμε τον Πάολο Κώστα και όταν ήταν εδώ στο κοινοβούλιο, βρισκόταν εδώ στο κτίριο, τον, τον, τον καρφώσαμε και έγραψε και εκείνος. Έχετε εδώ μέσα θαυμάσιες φωτογραφίες αναμνηστικές ε, από τη ζωή της Ούτα, την καριέρα της, ο κύριος Αλκαντράουι, Γκρόσ και η κυρία Μάισνερ και ο κύριος Κρέμερ, συγγνώμη, οι τρεις συντονιστές οι οποίοι έχουν μία πραγματικά ε, ε, λαμπρή έκφραση στο πρόσωπό τους κατά μια συνεδρίαση των συντονιστών τα έχουμε όλοι υπογράψει με διάφορα μηνύματα. Είναι ένα βιβλίο πραγματικά πολύτιμο το οποίο δείχνει ε, στην αγαπητή κυρία σε τι εκτίμηση την ε, έχουμε και πόσο, την, πόσο εξέχουσα εργασία έκανε και ο Μάικλ εδώ στο το ποδήλατο επάνω, ναι, θαυμάσια φωτογραφίες. Και θέλουμε να σα δώσουμε το βιβλιαράκι αυτό και μερικά άλλα δώρα τα οποία δίνουμε για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για το δύσκολο και λαμπρό έργο το οποίο επιτελέσατε. And of course Θα συμφωνείτε όλοι μαζί μου ότι η κυρία Κάσνιτς χρειάζεται δύο λεπτά για να απαντήσει. Δύο λεπτά μόνον αυστηρότατα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητή κύριε Βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την απόλυτη υποστήριξη που έλαβα τα τελευταία 7 χρόνια. Πραγματικά ήταν πολύ ενθαρρυντική όλη η υποστήριξη και ήταν εξαιρετική, θα έλεγα, αυτή η εμπειρία. Ελπίζω ως οικογένεια για θέματα μεταφορών να συνεχίσετε τις εργασίες και να περάσετε όλα τα σημαντικά πακέτα, ειδικά το πακέτο για τις αναρίες μεταφορές και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το έργο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του και για τον τρόπο με τον οποίο με υποστήριξε σε κάθε ε, θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Γιούτα και καλή τύχη και για τελευταία φορά θα... κάποιο κάποιος θέλει να μιλήσει. Ματ, έλα γρήγορα. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θέλουμε και εκ μέρους του ΕΛΚ και γραπτό ήδη έχουμε ευχαριστήσει, αλλά Θέλουμε και προφορικά να, ευχαριστήσουμε την κυρία Κάσνιτς γιατί συνήθως κάποιος ε, έχει τόσο μεγάλο χειροκρότημα όταν συνταξιοδοτείται. Αλλά τώρα η κυρία Κάσνιτς πηγαίνει στο Λουξεμβούργο. Μπορεί λοιπόν να μας ξαναεπισκεφθεί στις Βρυξέλλες. Η δουλειά της δεν ήταν πάντοτε η πιο απλή, ήταν ε, δύσκολο να επιτύχει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των ομάδων, αλλά η θέση της ε, ήταν πάντοτε εξαιρετική, ποτέ ε, δεν ήταν υποκειμενική και προσπάθησε πάντοτε να είναι όσο ουδέτερη και αντικειμενική μπορούσε. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και της ευχόμεθα κάθε επιτυχία στην περαιτέρω ε, ζωή της, ε, δεν ξέρω πού θα εργαστεί, αν θα εργαστεί στην πατρίδα της, αλλά ελπίζω να ξαναβρει το δρόμο στις Βρυξέλλες πίσω να μας επισκεφτεί. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ οι συντονιστές που θα πάρουν το λόγο να είναι σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ, Μπράιεν. Θα ήθελα κι εγώ εξ ονόματος ε, των συναδέλφων της δικής μου ομάδας να σας ευχαριστήσω ολόθερμα για το έργο σας. Δεν είναι καθόλου περίεργο που σας χειροκρότησαν ε, όρθιοι όλοι οι συνάδελφοι σήμερα εδώ. Είναι η απόδειξη της σκληρής δουλειάς που κάνατε τόσα χρόνια, διακριτικά, στα παρασκήνια, αλλά πάντοτε παρούσα. Ήσασταν ένα άτομο απόλυτης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας και δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο ότι οι εργασίες στην Επιτροπή μας έτρεξαν τόσο ομαλά τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε ολόθερμα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και κάθε επιτυχία και ικανοποίηση στις νέες σας δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ούτε όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος ε, την οποία είχε εσύ αυτά τα καθήκοντα στη γραμματεία ήταν μια εξαιρετική περίοδος. Μπορούσα πάντοτε να σε ρωτήσω σε κάθε ζήτημα το οποίο δεν καταλάβανα που ήταν μια, ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μένα. Ο Ματίας είπε ότι μπορεί να ξανάρθει στις Βρυξέλλες αλλά μπορούμε και εμείς να έρθουμε στο Λουξεμβούργο γιατί να μην έρθουμε εμείς να σε δούμε. Πολύ ωραία. Ο Πίτερ. Ναι, ούτε. Να σε ευχαριστήσω και εγώ. Ξέρετε, εμείς λέμε civil servants στα αγγλικά, είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά με την έννοια της υπηρεσίας του πολίτη. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπηρετήσετε τον πολίτη και ήταν η επιτομή αυτής της έννοιας. Πραγματικά υπηρετήσετε εξαιρετικά την Επιτροπή μας και θα πρέπει ουσιαστικά να σας δώσουν μια πλακέτα με χρυσά γράμματα με αυτόν τον τίτλο. Ήσασταν όχι απλά εξαιρετική δουλειά, ήσασταν και πολύ εγκάρδια και πολύ φιλική με όλους μας. Πιστεύω ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά, ήταν ήσασταν εξαιρετική υπάλληλο για το Κοινοβούλιο. Και εγώ ευχαριστώ την ε, Ούτα για την ε, στήριξη και την βοήθειά της σε όλα τα ζητήματα για μένα ήταν ιδιαίτερη χαρά ε, όταν ε, τρώγαμε το πρωινό μαζί, μαζί διότι είμαστε από γειτονικέ πόλεις και έτσι συνδεθήκαμε ιδιαίτερα. Η Ούτα αντιπροσωπεύει τις προσικές ε, αρχές του χαρακτήρα, οι οποίες είναι πάντοτε ακράδαντες, αξιόπιστες και αναλύωτες. Ε, και την ευχαριστώ από εκβάθους καρδίας. Σε ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ όλους. Όταν η κυρία Κάσνη θα φύγει, όλοι θα σηκωθείτε και θα... τώρα που θα φύγει, σηκωθήκατε και χειροκροτήσετε. Όταν εγώ θα φύγω, θα κλείσετε και την πόρτα πίσω μου και θα πείτε ουφ, Απαλλαχτήκαμε. Okay. Καλώς λοιπόν. Τώρα μπορώ να πω λοιπόν για τελευταία φορά. Παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας. Το λέει και η κυρία Κάσνιτς. Για τελευταία φορά θα μου πει το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ελέγξτε παρακαλώ τις κάρτες σας. Πέρα της ψηφοφορίας. Well, it is our lucky day the PPE are not won over as... Λοιπόν, δεν έχουν ένα επιπλέον ή του ΕΛΚ. Πώς και έτσι. Έκαναν φαίνεται μία προσπάθεια για την ούτε. Λοιπόν, Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες εδάφους ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδονησία. Τελική ψήφος μόνο. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ομόφωνα 39 υπέρ. Σας ευχαριστώ δεκτή. Ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Άβυσαρ. Άρθρο 2, σημείο 3, 51. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54 καταπίπτει. 54 ναι, καταπίπτει. Περνάμε τώρα στην 50 6 και 57 ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 56 και 57. Ξεκινάμε. Επαναλαμβάνω ψηφίζουμε την 56 και 57. Η 54 κατέπεσε. Συνεπώς. Ψηφίζουμε 56-57 και 58 του κυρίου Τέιλορ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτής, δεκτές μάλλον. 63 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση στο ΕΛΚ. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 60 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Για ησυχία λίγο. Ξέρω, φτάνουν οι γιορτές, αλλά λίγη ησυχία. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 62 έχει καταπέσει γιατί έγινε δεκτή 60. Περνάμε στην 73 Βαντάλεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 64 Τζίλε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 65 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 8 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 και 69 είναι ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 70 τώρα και 71. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 72 έχει αποσυρθεί. Η 74 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος λοιπόν. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 74. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 77 του Keith Taylor, είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 9 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 80 81 και 82 έχουν καταπέσει γιατί δεχθήκαμε την 9. Η επόμενη ψήφος είναι για την 79. Κατά διέρεστη ψήφος. Για μια στιγμή. Επειδή έγινε δεκτή η 9 θα ψηφίσουμε μόνο επί τη βάση μία ολιστικής, μόνο αυτό το κομμάτι. Είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84. Ποιοι είναι υπέρ, Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα για την 84. Ξεκινάμε. Υπάρχει μεγάλη διασπορά. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα επιπλέον. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. 85 και 86 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 και 88 ταυτόσημες. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 87 και 88. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Σοσιαλδημοκράτε πάντα έχουν ένα περισσότερο. Όχι. Ο κύριο Αλκαντράουι. Έχετε λάβει υπόψη σα το ότι έχουμε ένα μέλο επιπλέον και μπορούμε μάλλον 12 να ψηφίζουμε. Ναι. 12. Λοιπόν, προφανώ δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα και σα δίνουμε τη δυνατότητα να ψηφίζει ένα επιπλέον. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Ματιέ, θα στο κρατήσω αν λες ότι είστε πάντα υπέρ της μηχανής και όχι του Πρόεδρου. Πέρασε η ψηφοφορία και γίνεται δεκτή. 89 τώρα. Μάλιστα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 91. Keith Taylor. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 90 καταπίπτει. 92. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, έλεγχος για την 92, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται, ξεκάθαρα. 93. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 10 έχει καταπέσει. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 104 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή 104. 105. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 Βαντάλεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 111 που περιλαμβάνει την προφορική τροπολογία των πρασίνων. Έχετε διαφωνία για την προφορική. Τότε θα την ψηφίσουμε μαζί ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ή αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη 14. Όχι, για μια στιγμή. Στη 15. Στις 15 της Wills. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά τη συμβιβαστική με την 25. Αιτιολογική σκέψη 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 29-30 ταυτόσιμες ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική Β. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 32 του Κουν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32 γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά στις ψήφους. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, πρώτα θα ψηφίσουμε τη συμβιβαστική. Έχω την 34, αλλά έχει καταπέσει εφόσον γίνει δεκτή η συμβιβαστική C αγγλικό. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτήν. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική C αγγλικά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οπότε δεν χρειάζεται να επανέλθω στην 34. Συμβιβαστική D αγγλική. Και είναι υπέρ. Συγγνώμη, έχουμε εδώ ε, ψηφοφορία σε δύο κομμάτια. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι εξαιρώντας ε, και τα λοιπά. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Δεκτή λοιπόν η D αγγλικά. Η 36 τώρα, και η Taylor και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 έχει καταπέσει. Η 39. Η κυρία Τίκαου. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 41 Τέιλορ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ έχει καταπέσει μάλλον η 45 γιατί έχει γίνει δεκτή η 20 Περνάμε τώρα στη 48. Τσίλε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 Φώστα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κύριε Σάρισα. Καλώς. Λοιπόν, τώρα θα υπάρξουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές εδώ. Before we το επόμενο θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. So we have Mr. Krayenko, the Krayenko.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 αγαπητοί συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τον Διευθυντή, τον κύριο Τικρέαν. Και να σας πω ότι επειδή ο κύριος Μίθατε έχει μία εκδήλωση προς το Λουξεμβούργο, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα παρόν μαζί μας, όμως ο κύριος Δικρέν είναι ο εκπρόσωπός του, ο οποίος θα μας ε, κάνει μια παρουσίαση για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε όλες αυτές τις υπέροχες υποδομές που θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη, όμως που μόνο στα λόγια μένουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη. Ο κύριος Κόρτ έχει το λόγο. Παρακαλώ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 Δυστυχώ σε κάθε παρουσίαση ξεκινάμε μιλώντας για την παρούσα κρίση, καθώς η κρίση αυτή οδηγεί στη συρρήκνωση των δημόσιων δαπανών, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα μειώνει και τη δυνατότητα δανεισμού από πλευρά τραπεζών. Και δυστυχώς τα πρώτα πράγματα που την χάνουν και επίπτωση στις περικοπές είναι οι επενδύσεις και ξέρουμε ότι οι επενδύσεις είναι απαραίτητο για την μακροχρόνια ανάπτυξη, απασχόληση κτλ. Οπότε ελοχεύει ένα σημαντικό στον προκειμένου. Όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές ο δανεισμός είναι πολύ σημαντικό σημείο και βεβαίω σημαντικότατο στοιχείο προκειμένου είναι το μέσο των μεταφορών. Άρα το πρόβλημα είναι πώ θα διατηρήσουμε μία βιωσιμότητα στις μεταφορές και άρα βιώσιμη κινητικότητα μακροπρόθεσμα. Πρώτα απ' όλα να σας παραπέμψω στην Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε μέσα στο 2011 με την πρόσφατα αναθεωρηθήσα πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μετά από τη σχετική άσκηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ε, ένα νέο εργαλείο επενδύσεων, οπότε έχουμε όλα τα εργαλεία ήδη στη θέση τους, οπότε επιτρέψτε μου να σας πω με λίγα λόγια ποιοι είναι οι όροι επιτυχίας εναντί αυτής της κατάστασης. Μια πολύ σημαντική πτυχή κατά τη γνώμη μας είναι η επιλογή των σωστών προγραμμάτων. Η επιλογή των καλών προγραμμάτων, όχι οποιοδήποτε προγράμματος. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Εκεί θα δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεύτερο και σημαντικό, αλλά αφορά πιο πολύ εσάς και όχι τόσο εμάς, είναι ένα πολιτικό, διοικητικό, κανονιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να βρει σε χώρες που θα διέπει αυτές τις επενδύσεις και τρίτον τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Ο κ. Μπάρακ μετά θα πει πιο πολλά λόγια προκειμένου. Είναι η καλή προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων. Η τεχνική, χρηματοοικονομική, συμβουλευτική βοήθεια μπορεί να σας παραχθεί. Και τέταρτος όρος είναι Καλή όρη χρηματοδότησης. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω εντάχει τρία κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα, τι έχει κάνει έως σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μεταφορές. Ε, δεύτερον, τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και τρίτον, να διερευνήσουμε το πώς μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Τι έχει γίνει έως σήμερα. Τελευταία πενταετία, 2006-2010, Έχουμε δώσει 70 δισεκατομμύρια σε δάνει στον τομέα των μεταφορών, δηλαδή 14 δισεκατομμύρια ετησίως, εκ των οποίων 8 αφορούν τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα και αποτελούν ε, το 15% της χρηματοδότησης ε, συνολικά που έχει δοθεί στις μεταφορές. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο ρόλος της τράπεζας είναι κομβικό εν προκειμένου. Τι προσφέρουμε ελκυστικούς όρους σε αυτό το δανεισμό. Ο στόχος της τράπεζας δεν είναι το κέρδος, γι' αυτό είναι ιδιαίτερο χαρακτήρα τράπεζα. Ε, οι στόχοι που επιδιώκει είναι ευρωπαϊκοί στόχοι, έπειτα. μακροπρόθεσμα, γιατί θα επανέλθω και μετά σε αυτό το θέμα το οποίο είναι κομβικό για τις υποδομές, είναι να δώσουμε ένα μεικτό εργαλείο στο οποίο εντάσσουμε δάνεια και επιχορηγήσεις και θα επανέλθω και σε αυτό ε, σε λίγο. Αυτά κάναμε τα τελευταία χρόνια και ε, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, τι πρέπει να γίνει μετά. Η Λευκή Βίβλος της Κομισιόν για τις μεταφορές δίνει κάποια πραγματικά στοιχεία που εκπλήσουν 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στις μεταφορές, στις υποδομές μεταφορές για την επόμενη 20 εκ των οποίων 550 δισεκατομμύρια για την ευρωπαϊκά δίκτυα έως το 2020. Τεράστια τα ποσά παρά τα αυτά. Αν τα συγκρίνουμε το τι έχει γίνει έως τώρα, τα τελευταία δηλαδή χρόνια, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο εκπληκτικά αυτά τα στοιχεία, γιατί για παράδειγμα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έως το 2% του ΑΕΠ αφορά αυτές τις επενδύσεις, ενώ στα παλαιά κρατημέλη είναι το ίμιση αυτό το ποσοστό. Άρα βλέπετε πώς ουσιαστικά φτάνουν το μέσο όρο τα νέα κρατημέλη και αυτό το 1,5 εκατομμύρια ευρώ κατανοείτε τι σημαίνει για κάθε έτος αυτής της 20 και είναι ουσιαστικά το 0,5% του ΑΕΠ. Άρα είναι πολύ λιγότερο από ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Παρά τα αυτά είναι μια τεράστια πρόκληση σε μια εποχή κρίσης. Θα περάσω τώρα στο πώς θα εξεύρουμε τους πόρους για να γίνουν αυτές τις επενδύσεις. Πώς θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που συρρυκνώνουν τα δημόσια οικονομικά στοιχεία και άρα επηρεάζουν ε, ταυτόχρονα και τον τραπεζικό δανεισμό. Σίγουρα θα έχετε ακούσει την έννοια των χρηματοπιστωτικών εργαλείων υπό την έννοια της νέας προσέγγισης. Δηλαδή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός συγγνώμη, από κοινού με τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να προσελκύσουν ιδιωτικά κονδύλια. Στην διαφάνεια υπαριθμών 6, που την, σας τη δείχνω πριν την διαφάνεια 5, βλέπετε ότι θα συνεχίσουν να πετούνται επιχορηγήσεις, όπως θα συνεχίσουν να πετούνται και δάνεια. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο εργαλεία, καθώς πάντοτε έχουμε ως γνώμονα ε, σαφώς οικονομικά δικαιολογημένα, τεκμηριωμένα ε, ε, προγράμματα δηλαδή που θα έχουν ένα όφελος για όλη την κοινωνία. Λοιπόν, αν αυτά τα προγράμματα δεν μπορούν να καλυφθούν από δάνεια, θα πρέπει να υπάρχουν και επιχορηγήσεις και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα μείγμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνεται κατασπατάληση πόρων, θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο μείγμα χρηματοδότησης ώστε να δοθούν πιο πολλά κονδύλια από ότι μια απλή επιχορήγηση, γιατί υπάρχει μόχλευση της ε, επιχορήγησης επί του δανείου και θα αναφέρω ως παράδειγμα μετά τα ομόλογα έργων. Και άρα εκεί χρησιμοποιείται και ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ε, τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν θέλω να πω πιο πολλά για την εμπειρία που έχουμε εμείς στην τράπεζα από τα PPP, τις εταιρικές σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εδώ ο συνάδελφος ε, μετά θα σας πει πιο πολλά γι' αυτό. Να πάω κατευθείαν στο παράδειγμα των ομολόγων έργων, τα project bonds. Είναι ένα μόνο παράδειγμα τέτοιων εργαλείων, χρηματοπιστωτικών εργαλείων που έχουμε καλό είναι να αφιερώσουμε ένα λεπτό από το χρόνο μας για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτή η έννοια. Αυτά τα ομόλογα έργα δεν είναι ευρωομόλογα. Δεν είναι ευρωομόλογα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη σύγχυση μεταξύ των δύο. Δεν κρίνω κανένα από τα δύο, αλλά τα ομόλογα έργων χορηγούνται, εκδίδονται από τον ιδιωτικό τομέα, από την εταιρεία που φέρει πέρα στο project. Αν πάτε στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε δεν ξέρω αν το διαβάζετε, στη διαφάνεια. Εδώ ε, σκεγγραφείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Βλέπετε το SPV στην αριστερή στήλη είναι το κόστος του project. Για παράδειγμα, μια οδική αρτηρία. Πάτε μετά στην δεξιά στήλη και βλέπετε το κεφάλαιο που πέφτει στο project και χρειάζονται ομόλογα επί του έργου, επί του project, ε, και χρηματοδοτείται αυτό το μέρος του έργου με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσελκυστούν όλα τα κονδύλια που απαιτούνται για την ε, ε, ολοκλήρωση, αν θέλετε, του project, χρειάζεται ενίσχυση της ε, πίστοσης, δηλαδή κάποιος πρέπει να αναλάβει έναν υψηλότερο κίνδυνο αυτό το βλέπετε στο μεσαίο κομμάτι της δεξιάς στήλης, για να μπορέσει αυτό τελικά το ομόλογο να επιτρέψει να το αγοράσουν οι ιδιώτες επενδυτές. Και εκεί χρησιμοποιείται και ο ευρωπαϊκός προπολογισμός σε ένα ποσοστό για να καλύψει το πρώτο ε, κομμάτι που, ε, έχει, που λείπει το ενδιαφέρον σε αυτό το σχέδιο... Α, συγγνώμη, χάσαμε τη διαφάνεια, λέει ο μιλητής, αλλά απαιτείται μια μικρή συμβόλαιο του προλογισμού 4 δις εξαρτάται. Αν έχουμε ομόλογα 100 εκατομμυρίων, με 4 εκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, μπορείτε να έχετε 20 εκατομμύρια από την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξετε σε ομόλογα 100 εκατομμυρίων. 4 εκατομμύρια από τον υπολογισμό, 20 εκατομμύρια από την Τράπεζα Επενδύσεων, καταλήγουμε στο μόλογο 100 εκατομμύριων. Και έτσι θα καλυφθεί η ανάγκη ε, επένδυση 150 εκατομμύριων. Βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται η μόχλευση. Από 4 εκατομμύρια ξεκινάτε από τον υπολογισμό και καταλήγετε να καλύπτει μια επένδυση 150 εκατομμυρίων. Να, ε, η αξία αυτής της προσέγγισης. Ένα μόνο παράδειγμα είναι τα ομόλογα έργων. Υπάρχουν και πολλά άλλα ε, παραδείγματα άλλου είδους εργαλεία κεφαλαίων, αλλά αυτό το μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στον τομέα των μεταφορών. Σα παραπέμπω και σε πέντε εργαλείο όπω το LGTT για τι ε, μεταφορέ που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν. Θέλω να πω όμω ότι η χρηματοδότηση δεν αρκεί. Πέρα από την χρηματοδότηση, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η προετοιμασία του έργου ε, του προγράμματο. Και εδώ έχουμε στενή συνεργασία με την Κομισιόν για να προετοιμάσουμε αυτό το κομμάτι και επ' αυτό θα τοποθετηθεί ο κύριος Μπάρεξ λίγο ώστε να υπάρξει καλύτερη επιλογή των project, να υπάρξει καλύτερη ιεράρχηση των ενδιαφέροντος και υπάρχει και το Jasper που θεωρητικά τα θεωρητικά ταμεία, το Jessica, το EPEC που θα δούμε σε λίγο και πολλά άλλα τέτοια εργαλεία. Και να κλείσω επί του θέματος λέγοντας, όπως είπα, εν είδη εμείς στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πιστεύουμε ότι η απέντηση είναι θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Και αυτό ισχύει απόλυτα στις υποδομές των μεταφορών. Και μέσα στα πλαίσια μιας κρίσης που οδηγεί σε συρρήκνωση των προϋπολογισμών, των δημόσιων προπολογισμών και των τραπεζικών ε, πιστώσεων, να ένα τρόπο. για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να γεφυρώσουμε αν το χάσμα και να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε τι προτεραιότητε της Ένωσης με απόλυτη λογοδοσία προ τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους εργαλεία όπως είναι τα ομόλογα έργα θα πραγματικά θα δημιουργήσουν μόχλευση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και ταυτόχρονα θα επιτρέψουν και σε εμά την τράπεζα να παρέχουν περισσότερες ε, επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ντεκρέν και θα ε, συνεχίσω με τον κύριο Μπάρετ και μετά μπορούμε να κάνουμε μια γενική συζήτηση. Okay, Mr. Barrett. Λοιπόν, κύριε Μπάρετ, είστε επόμενο. ήταν ο πρώην διευθυντή της ECB για την ε, βόρειο-δυτική Ευρώπη, κρίσιμο σημείο η νότιο-δυτική Ευρώπη και ό,τι έχει κάνει ο κύριο Μπάρετ είναι λίγο σημαντικό. Και είναι τώρα εμπειρογνώμων σε ό,τι αφορά τα κοινά προγράμματα δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, τα περίφημα 3P. PPP και του δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να σας κάνω την παρουσίασή μου σήμερα το πρωί και αυτό που ε, θα προσπαθήσω να κάνω είναι να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία κλειδιά. Για να ε, μπορέσω να σας ε, παρουσιάσω ένα μήνυμα διότι πολλές φορές αυτά τα κοινά προγράμματα δημόσιο ιδιωτικού τομέα είναι συγκεχημένα και πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς τι αντιπροσωπεύουν. Καταρχάς, μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα και στο, μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο υπάρχει μία εδρεωμένη μεθοδολογία συζήτησης ε, ή χειρισμού, αν θέλετε, των προγραμμάτων αυτών, των PPP άπτεται του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, καθορίζει λεπτομερώς ποια είναι τα όρια, οριοθετεί δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των δύο τομέων και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και των εταίρων. Στην ουσία αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο για την διαχείριση δημοσίων επενδύσεων. Ένα επιπλέον πρόσθετο εργαλείο για να βοηθήσει την επίτευξη των στόχων του δημόσιου τομέα. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε τι έχει επιτευχθεί στον όλο τον τομέα των ε, δημοσίων ιδιωτικών επενδύσεων, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο επενδύσεων. Ήδη το οποίο έχει γίνει στα πλαίσια αυτά. Εάν δείτε τα στοιχεία, 30 δις ε, επενδύσεις ετησίως και τα πιο αδύναμα έτη, το χαμηλότερο ας πούμε, ήταν ε, το ίμιση αυτού του ποσού ή λίγο λιγότερο από το ίμιση. Υπάρχει λοιπόν ε, μια ευελιξία όσον αφορά τη ζήτηση αυτού του εργαλείου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη των στόχων των δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, αν κοιτάξετε την γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων αυτών, στην αρχή ε, τα κοινά έργα δημοσίου ιδιωτικού τομέα ε, υποστηρίχθηκαν πλήρως από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο αυτό ε, μοντέλο ισχύει ακόμα. Το 2010 η Ισπανία ήταν η βασική αγορά μέσα στην οποία κινήθηκαν τα, τα έργα αυτά ε, με τη μορφή του PPP. Εν συνεχεία το, το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο μετακινήθηκε από τα μεγάλα έργα, επενδυτικά έργα δημόσιου ιδιωτικού φορέα, σε κοινοπραξίες δηλαδή, σε μικρότερα. Και το 2011 φέτος η Γαλλία θα είναι η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις κοινοπραξίες διότι ο δημόσιος φορέας στήριξε ιδιαίτερα την ιδέα αυτή και τον τύπο αυτών των ε, κοινοπραξιών. Η Γαλλία λοιπόν θα είναι επικεφαλής. Φέτος ε, είμαστε τώρα σε μια νέα θέση, κατέχουμε μια νέα θέση όταν εξετάζουμε τις κοινοπραξίες αυτές, όχι μόνο στα μεγέθη αλλά ε, πώς ε, χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν δείτε τις βασικές οικονομίες μέσα στην Ένωση, θα σημειώσετε ότι το εύρος των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι, κυμαίνεται από 2% στη Γερμανία μέχρι περίπου 6% στην Πορτογαλία ως ποσοστό του ΑΕΠ με μέσο όρο το 2008. Εδώ δείχνει λοιπόν την, το μέγεθος της οικονομίας και τις επιλογές που κάνουν οι κυβερνήσεις στο κατά πόσο θα χρησιμοποιούσαν αυτές τις κοινοπραξίες και κατά πόσο έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Για τους στόχους τους, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Πορτογαλία και όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής, η Γερμανία και η Πολωνία δείχνουν ότι υπερέχουν του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά τα μεγέθη και τη χρήση των ε, κοινοπραξιών αυτών, ενώ άλλες, οι υπόλοιπες χώρες υπολείπονται. Εάν τώρα ε, εξετάσουμε τους ε, τομείς όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι επενδύσεις, ο τομέας των μεταφορών ήταν πάντοτε πολύ βασικός. Ε, βεβαίως και η παιδεία και οι υπηρεσίες υγείας και άλλοι τομείς, αλλά οι μεταφορές κατέχουν ένα σημαντικότατο, μη σημαντικότατη θέση σε αυτές τις επενδύσεις. Εν συνεχεία, γιατί χρησιμοποιούνται αυτές οι κοινοπαξίες. Χρησιμοποιούνται διότι αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέβρεση ε, επιπλέον πόρων και εμπειρογνωμοσύνης που θα μπορέσουν να στηρίξουν ε, τη στοχοθέτηση των δημοσίων τομέων. Σας είπα ότι ήδη η κοινότητα έχει ταυτοποιήσει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες. Ξέρουμε ότι οι κοινοπραξίες αυτές είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί μόνο στις συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν είναι μία λύση ευρέως φάσματος, αλλά εν πάση περιπτώσει με τις παρούσες συνθήκες ούτε οι αγορές ούτε οι εθνικοί προϋπολογισμοί μπορούν να εκπληρώσουν τα, τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση. Πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνα τους υπάρχοντες δημοσιονομικούς ε, πόρους. Και εδώ ακριβώ υπησέρχεται ο ρόλο αυτών των κοινοπραξιών, διότι επιτρέπει στο δημόσιο τομέα να βρει, δημόσιες, να βρει κονδύλια, να βρει πιστώσεις εκτός κοινοτικού προϋπολογισμού, διευκολύνει τη χρηματοδότηση με τις, από τις τράπεζες και τις κεφαλαιογορές και επιτρέπει τις επενδύσεις, να, τον προγραμματισμό των επενδύσεων να γίνει με προσεκτικό τρόπο. Οπότε, όταν μιλάμε για τις ε, κοινοπραξίες αυτές αναφερόμαστε σε ένα λίαν στρατηγικό δημοσιονομικό εργαλείο το οποίο προσφέρει πρόσθετη αξία και διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση των πόρων, των δημοσιονομικών πόρων. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ότι οι κοινοπραξίες αυτές είναι εκτός ισολογισμού αυτό πλέον δεν ισχύει. Και επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat για τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα δεν το υποστηρίζουν και δεύτερον επειδή χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στην δημοσιονομική διαχείριση όλων των οικονομικών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ε, δανειοδότηση κατά 2 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ε, των, κοινο, των κοινοπρακτικών αυτών προγραμμάτων. Περίπου το 50%, το 50% Θέλω να τονίσω, συγγνώμη, περίπου το 15% των προγραμμάτων μας έχει χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Ε, τα, η χρηματοδότηση των PPP είναι μεν ένα εργαλείο, αλλά όχι το μόνο για την εφαρμογή των δημοσίων στόχων. Όμως είναι λογικό να πούμε ότι επειδή πολλές χώρες έχουν αυτά τα προγράμματα, πρέπει να καταλάβουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και γι' αυτό υπάρχει ακριβώς αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, το EPEC. Ε, ο ρόλος αυτού του κέντρου είναι η διανομή της τεχνογνωσίας, η διευκόλυνση των δημοσίων αρχών να διαχειριστούν ε, τα κοινοπρακτικά αυτά προγράμματα, η, η ενημέρωση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το επιτύχαμε επικεντρώνοντας την προσοχή μας περισσότερο στην ανάπτυξη του δυναμικού, ε, στην ε, παροχή ε, στήριξης στρατηγικών πολιτικών και στην ανάλυση και μελέτη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Η εφαρμογή λοιπόν των βέλτιστων της βέλτιστης έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την καλή χρήση αυτού του εργαλείου. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναγνωρίζει σαφέστατα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνεργασίας με τις εθνικές αρχές για να αλληλοσυμπληρώνονται τα ωφέλη τα οποία έχουν και οι δύο πλευρές και τα πλεονεκτήματα. Αυτό το κάνουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία όχι μόνο προσφέροντας ε, χρηματοδότηση αλλά προσφέροντας και εμπειρογνωμοσύνη και ε, συμβουλές σε δημόσια έργα. Σας ανέφερα ήδη ορισμένα παραδείγματα. Υπάρχει το πρόγραμμα Jessica επίσης το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, αστική ανάπτυξη αστικών περιοχών και χρησιμοποιεί κονδύλια του Διαρθρωτικού Ταμείου και το πρόγραμμα Jaspers, το οποίο αντιπροσωπεύει είναι ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση του, των έργων του Διαρθρωτικού Ταμείου, Ειδήσεων των τομέα μεταφορών. Έχουν ε, μια πάρα πολύ καλή ε, ανάπτυξη αυτά τα προγράμματα και πιστεύω ότι αρκετά μέλη αυτού του σώματος έχουν εμπειρία από τα δύο αυτά προγράμματα και πόσο καλά έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα. Αυτά, Πρόεδρε, είχα να πω ε, σε μια γενική παρουσίαση του θέματος και είμαι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάρτ και κύριε Ντεκρέιν και έχω τους ομιλητές. Um, Όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο παρακαλώ να μας το υποδείξουν. Ο κύριος Γκρός πρώτα απ' όλα. vielen Dank, Herr Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Σήμερα θέλω να περιοριστώ στις τεχνικές χρηματοδότησης, γενικά στο, στην οικονομική πτυχή. Ε, είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά τα οποία μας είπατε τα χειρίζεστε με μεγάλη επιτυχία. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση αφορά το εξής πόσο πιστεύετε ότι ε, η οικονομική υποδομή ενός έργου είναι εφικτή, πόσο αξιόπιστη είναι η οικονομική έκθεση για ένα έργο ε, και τι στοιχεία χρειάζονται για να μπορέσει η Κομισιό να βασιστεί σε αξιόπιστα, σε μια αξιόπιστη οικονομική διαχείριση του προγράμματος. Δεύτερον, η οι χώρες που προετοιμάζονται για να, στη χρήση αυτών των κοινοπραξιών, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή αυτό το εργαλείο, έχουν προχωρήσει, έχουν ξεκινήσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς ε, για την εκτέλεση ε, τέτοιων κοινοπρακτικών έργων. Έχετε γνώση για τη συνεργασία κοινοπραξιών υπό το πλαίσιο αυτών των ε, τριών του PPP, αυτής της ε, αρχής. Και όσον αφορά τώρα τα ομόλογα έργων, είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον των σιδηροδρόμων. Και είχαμε συζητήσει τι είδος ε, έσοδα μπορούν να έχουν οι ανεξάρτητοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην λειτουργία των σιδηροδρόμων. Παραδείγματο χάρη αυτοί οι εταιρείε στις οποίες ανήκουν οι γραμμές, οι, οι σηματοδοτήσεις κλπ. Ε, είναι για σας σημαντικό σημαντικό να έχετε στοιχεία και πώς θα διαχειριστείτε τις απαιτήσει προσόδων των εταιριών, των ανεξαρτήτων αυτών εταιριών για να κρίνετε αν μπορούν να ενταχθούν στο, στις, στις κοινοπρακτικές αυτές ε, επιχειρήσεις και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να, και να κρίνετε τι κονδύλια με τι κονδύλια μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και τέλος, όσον αφορά αυτά τα, τις κοινοπραξίες, δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Ε, τα έργα τα οποία έχουν οικονομικό όφελος, όπου δηλαδή οι πρόσοδοι, τα έσοδα ή το κέρδος ε, έχει ληφθεί υπόψη στην όλη διαχείριση, διαφέρουν ασφαλώς από έργα τα οποία δεν έχουν ε, κέρδος ή δεν σημειώνουν, δεν έχουν έσοδα. Ποιο λοιπόν, ποια λοιπόν αρχή σας ενδιαφέρει περισσότερο, θα εξετάσετε τα στοιχεία των απο, της απόδοσης των προσόδων για να κρίνετε ποια έργα θα εγκρίνετε ή όχι. Ο πρόεδρος, θα ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις για να δώσουμε μετά την ευκαιρία σε απαντήσεις. Ο κ. Αλ Καντράουι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σχετικά με τα project bonds αν έχω καταλάβει καλά, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και η δυνατότητα βελτίωσης του χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων ομολόγων, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτών επενδυτών. Διερωτώ με πάντως σε αυτή τη φάση ποια είναι αξιοπιστία αυτών των συστημάτων αξιολόγησης βέβαια γιατί τα συστήματα αξιολόγησης τα οποία είναι γνωστά μέχρι τώρα στην ουσία δημιουργούν δυσκολία στην κυκλοφορία των συγκεκριμένων αυτών ευρωπαϊκών ομολόγων. Και διαρωτώ με αν οι αρχές ε, ακριβώς λόγω αυτών των ομολόγων από την άλλη μειώσουν τις λεγόμενες διαρθρωτικές επενδυτικές δημόσιε προσπάθειε τις οποίες κάνουν μέχρι τώρα. Και έτσι σε αυτή την περίπτωση οι σιδηρόδρομοι θα καταδικαστούν σε εισαγωγικά ε, στην χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών μέσων καινοτόμων όπως τα project bonds. και τα χρήματα σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι προφανώς επαρκή. Κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το κόστος της ανανέωσης των υποδομών και ελπίζω να καταλάβατε τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση που δημιουργείται φαίνεται να είναι σχετικά περίπλοκη. Θα δείτε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι κίνδυνοι ε, πέφτουν περισσότερο και τους αναλαμβάνουν περισσότερο ε, οι φορείς του δημοσίου, ενώ οι ιδιωτικοί φορείς πάντα έχουν κάποιες μορφές εγγυήσεων για τη μία απώλεια των επενδύσεών τους. Οπότε τι επιλογές έχουμε εδώ, είτε να μην κάνουμε καθόλου επενδύσεις, είτε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις σχετικά πιο ακριβές για το φορολογούμενο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες επιπτώσεων σαν παράδειγμα ανάμεσα στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 100% από το δημόσιο και σε προγράμματα τα οποία οφείλονται στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, τα PPS. Και ποια είναι η κατανομή του κόστους ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Έχουν ήδη τεθεί αρκετές ερωτήσεις, δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ πάρα πολύ ώρα. Να πω κάτι μόνο προς τον κύριο Ντεκρέγιον Κούρ. Διαρωτώ με τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε και τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν και από τις νέες μορφές ομολόγων. Δύο ερωτήσεις. Ε, τα πιλωτικά προγράμματα πότε θα ξεκινήσουν πρώτον και τι μέγεθος θα έχουν δεύτερον. Όλη Ρεν αναφέρθηκε σε μια δυνατότητα για τις μεταφορές ε, για 4 δις, αν κατάλαβα καλά. Επιπλέον είναι αυτά τα 4 δις. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τι ρόλο θα παίξει σε σχέση και τι ποσοστό θα καλύψει σε σχέση με αυτά τα, με αυτά τα ποσά. Ξέρουμε ότι τα ποσά αυτά δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, παρόλα αυτά φαίνονται αρκετά ελκυστικά. Και στις ε, σημερινές συνθήκες, οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες, ε, ίσως κάποιοι να αντιδράσουν και να θεωρήσουν ότι είναι υπερβολικά υψηλά. Υπάρχουν επίσης χώρες όπως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία όπου ε, πρέπει να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι ιδιώτες ε, ε, επενδυτές γιατί το δημόσιο από πλευράς του παίζει πλήρως το ρόλο τον οποίο καλείται να παίξει. Κυρία Φώστα, ευχαριστώ Πρόεδρε για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο αλλά κάνατε μια παρουσίαση αρκετά κατανοητή. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να κυκλοφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να υπεραπλουστεύει κανείς την κατάσταση, ε, πώς πιστεύετε ε, για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Έχουν υπάρξει δανειοδοτήσεις, αρκετά χρήματα έχουν κυκλοφορήσει, ομόλογα έχουν κυκλοφορήσει και θα κυκλοφορήσουν. Πώς ελέγχετε εσείς τη σωστή τους χρήση. και πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ελέγχει τα χρήματα τα οποία διαθέτει σε σχέση με τη σωστή τους κατάληξη και χρήση. Απαιτείται και πολιτική παρέμβαση φοβάμαι πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρω πώς θα πετύχετε κάτι τέτοιο. Εάν πράγματι θέλετε, θέλει κάποιος να πάρει ένα δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και απορριφθεί η αίτησή του. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός ε, για να μπορέσει κανείς να εφεσιβάλει την συγκεκριμένη απόφαση. Έχουμε δει εξαιρετικά προγράμματα τα οποία να ολοκληρώνονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινοτικά χρήματα και είδαμε όμως και αρκετά προγράμματα στα οποία τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου δεν πήγαν και σε πολύ καλούς στόχους. Είδα πολλά, τα, τα μάτια μου είδαν πολλά όταν ήμουνα στα ΑΚΕΑ, ας πούμε, στην πρώτη κοινοβουλευτική περίοδο που υπηρέτησα. Υπάρχουν επίσης και οι μικτές ε, τεχνολογικές πρωτοβουλίες και στον τομέα των ουρανών και της απομόλυνσης ε, σε σχέση με τις εκπομπές καυσαερίων και σε σχέση με τις φαρμακευτικές ουσίες είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στην βιομηχανία όταν αυτό το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει και είχαν υπάρξει πάρα πολλοί φόβοι γιατί η βιομηχανία είχε κάνει πολλές επενδύσεις τις οποίες δεν έβλεπε να πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό το γύρο ο κύριος Κράμερ για τρία λεπτά. Στη Γερμανία είναι σαφές ότι χρειάστηκαν για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο σημείο το οποίο είμαστε σήμερα πάρα πολλές επενδύσεις. Είχαμε πει πριν από αρκετά χρόνια ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες επενδύσεις. Οι επενδύσεις θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε παντού, να κάνουμε δημόσια έργα παντού, αλλά η απόδοση φυσικά από τις συγκεκριμένες αυτές ενέργειες ε, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 15 χρόνια. Είχαμε συζητήσει και με τους ελβετικούς ιδιοδρόμους, για, την, για τον συνδυασμό και τον συντονισμό αυτών των επενδυτικών και ε, προσπαθειών αποκατάστασης των υποδομών κυρίως και φάνηκε ότι είχαμε αρκετά προβλήματα. Είχαμε προβλέψει ένα κοινό τέτοιο πρόγραμμα για τον άξονα Λιών του Όρινο όπως επίσης και Βασιλεία Μπρέμεν. Εκεί ε, είδαμε ότι για να είναι αποδοτικά τα προγράμματα αυτά θα έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Το είδαμε και σε μικρότερες κλίμακες, στη σύνδεση σαν παράδειγμα Μπρέσλαου-Βερολίνου. Ε, προχωρήσαμε από την άλλη, θα πρέπει να υπάρξουν ας πούμε και διζελομηχανές ή ηλεκτροκίνητες μηχανές, τις οποίες ποιος θα τις πληρώσει αυτές για να κερδίσουμε έστω και αυτή τη μισή ώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο συνδυασμός με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητος. Ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος επενδύει δεν μπορεί να περιμένει 40 χρόνια για να πάρει τα χρήματα του πίσω. Αν κάνουμε τέτοιου είδους υπολογισμούς δεν χρειαζόμαστε το ιδιωτικό σε εισαγωγικά χρήμα. Το δημόσιο μπορεί μόνο του να δει τόσο μακροπρόθεσμα, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί. Στη Γερμανία όταν ας πούμε ε, χτίζουμε καινούριου αυτοκινητοδρόμους τους κάνουμε με εκχώρηση της χρήσης τους από τις εταιρείες οι οποίες τους χτίζουν. Και αυτή η εκχώρηση χρήσης και εκμετάλλευση αυτών των αυτοκινητοδρόμων είναι ε, τουλάχιστον, έχει τουλάχιστον διάρκεια 20 ετή. Λοιπόν, οι εμπειρίες ε, τις οποίες είχαμε, ε, είδαμε ότι ο συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι κάτι το εφικτό. Θυμάστε ε, τι είχε πει η Θάτσερ κάποτε για την σύραγγα, την σύραγγα ότι θα, για τη, της ότι θα διχτήσουμε μένα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πληρώσει το κράτος για αυτού του είδους την επένδυση. Η αλήθεια είναι ότι δεν πλήρωσε το κράτος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας έχασε πάρα πάρα πολλά χρήματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς το χρέος το οποίο έχουμε ε, για επενδύσεις αλλά και το χρέος το οποίο κουβαλάμε σαν κράτη να το ρίχνουμε στις πλάτες του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, κύριε Ντεκβενιακού ξεκινήστε και μετά ο κύριος Μπάρετ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που καταδεικνύουν τον ενδιαφέρον της Επιτροπής σας για το θέμα. Κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Πολύ εξημών θέσατε το ζήτημα της διαδικασία επιλογής των προγραμμάτων. Δηλαδή πώς εντοπίζονται, πώς επιλέγονται τα προγράμματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι η επιλογή δεν γίνεται με πολιτικό κριτήριο, αλλά η επιλογή γίνεται με γνώμονα μια συγκεκριμένη πολιτική. Ε, είναι διαφορετικό αυτό που λέω. Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Η πολιτική της Ένωσης έχει καθοριστεί σε μια σειρά εγγράφων που ανέφερα πριν στην παρουσίαση μου. Οπότε να γνωρίζετε, παρακαλώ, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απασχολεί περίπου 280 επιρογνώμονες ειδικού σε αυτά τα θέματα, όπως είναι μηχανολόγοι, οικονομολόγοι, εξειδικευμένοι άνθρωποι σε όλους τους τομείς, μεταξύ αυτών των τομέα των μεταφορών, όπου αξιολογούν λεπτομερώς κάθε πρόγραμμα. Πηγαίνουν επί και αξιολογούν το, ε, την πρόταση, την οικονομική του αξία, την ε, οικονομική αξία και το όφελος για την κοινωνία γέννη, τον τεχνικό σχεδιασμό, κατά πόσον οι προδιαγραφές του συνάδουν με τις καλές πρακτικές, ελέγχουν βεβαίως την οικονομική του βιωσιμότητα. Αυτή τη στιγμή ζητείται ένα δάνειο. Ε, τον ε, αντίκτυπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, όλα λοιπόν αυτά συνεξετάζονται από πλευράς μας και όχι από κάποιον τρίτο. Και η δική μας εμπειρία, όπως ε, έχει χτιστεί σε άλλους τομείς και σε άλλες χώρες, πάντοτε ε, μας βοηθά στην επιλογή. Οπότε, ελέγχουμε κατά πόσον η κάθε πρόταση επιρετεί την γενικότερη πολιτική της Ένωσης και κατά πόσον θα έχει αυτή την απόδοση. Τώρα, το μέγεθος η τράπεζα μας έχει την έδρα και στο Λουξεμβούργο, έχει 2.000 περίπου υπαλλήλου, οπότε δεν μπορεί να ελέγξει ε, και τις τελευταίες λεπτομέρειες μικρών προγραμμάτων. Οπότε έχουμε ένα σύστημα όπου ε, κάποιοι ε, χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές θα ελέγξουν τα μικρά προγράμματα. Εμείς βεβαίως ελέγχουμε τα μεγάλα προγράμματα, δηλαδή αυτά που είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ πέρα από το μέγεθος, θέσατε και, κύριε Μέσνερ, ένα άλλο ερώτημα για τα ομόλογα έργων, για τα project bonds. Είναι ένα εργαλείο τα project bonds που έχει ως σκοπό στο επόμενο πολιτές μεσονοκό πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Όπως ορθά μου είπατε, αυτή τη υπάρχει μια πρόταση από την Κομισιόν να κάνει ένα πιλωτικό project, το οποίο έχετε λάβει και εσείς ως πρόταση να συζητήσετε και θα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά κυρίως για τις μεταφορές. Και τα τέσσερα δις που αναφέρατε εσείς αφορούν την πιλωτική περίοδο, δηλαδή μόλις εσείς το εγκρίνετε, έτσι, το στομότερο δυνατόν, προς όφελό σας είναι. Γιατί ε, η πιλωτική αυτή περίοδος θα τρέξει στο 2013. Έπειτα ο κύριος Γκρός έθεσε ένα άλλο ερώτημα είπατε γιατί να χρησιμοποιούνται δάνεια, επιχορηγήσεις και γιατί ε, χρησιμοποιούνται και μεικτά εργαλεία. Να σας παραπέμψω πάλι στην διαφάνεια υπαριθμών 7. Ίσως την έτρεξα πολύ γρήγορα, γιατί εκεί σας δίνω το πλαίσιο για αυτή την προσέγγιση που επιλέξαμε. Δηλαδή, αν ένα project... Δεν μιλάμε για τα project που δεν είναι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καλό project, όπως το περιέγραψα πριν, και θα έχει ε, υψηλή οικονομική απόδοση ή πολύ χαμηλή αρνητική απόδοση, Μιλώ για τον επενδυτή, τον ε, ε εκάστοτε επενδυτή λοιπόν. Αν είναι χαμηλό ο κίνδυνο και υψηλό το κέρδο, τότε δεν χρειάζεται να μπει κανένα θεσμικό ε, παράγοντα. Η αγορά θα το καλύψει μόνο. Αν όμω είναι χαμηλή οικονομική απόδοση, θα υπάρξει ζημία ή υπάρξει πολύ ψηλό κίνδυνο. Εκεί, ναι, θα πρέπει να λειτουργήσει με επιχορηγήσει, όπω είναι τα διοσυνοριακά προγράμματα, τα διοσυνοριακά project πολύ συχνά πέφτουν σε αυτήν την κατηγορία, γιατί εκεί ο ιδιώτη επενδυτή διστάζει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, οπότε χρειάζονται επιχορηγήσει. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μέση ζώνη, όπου είναι χαμηλό το οικονομικό κόστο και υψηλό ο κίνδυνο με κάποιε επιχορηγήσει μπορεί να μοχλεύσει ε, δάνειο από την ε, Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να ξεκινήσει αυτό και να προσελκύσει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η προσέγγιση που επιλέξαμε για αυτή την κατηγορία. Στην κυρία Φώστερ να πω συμφωνώ και επισημαίνω και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν λαμβάνει και δεν διαχειρίζεται χρήματα φορολογουμένων. Τα δάνεια που εμείς χορηγούμε προέρχονται από δανεισμό από τις χρηματαγορές. Η δική μας τράπεζα είναι μια τις μεγαλύτερους οργανισμούς έκδοσης ομολόγων και άρα εμείς ουσιαστικά αντιλούμε χρήματα από τις χρηματαγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε σημασία στον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δάνεια και αποπληρώνονται. Το αντίθετο, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις, το δάνειο όταν το δίνεις, θέλεις ο απόλυτα να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Άρα υπάρχει πολύ αυστηρή παρακολούθηση, ενδελεχής παρακολούθηση για την υλοποίηση του project, αλλά και εκ των προτέρων κατά πόσο θα έχει τη δυνατότητα να αποπληρωθεί το δάνειο. Και είμαστε περήφανοι για τη δίκαση που ακολουθούμε και πιστεύουμε ότι αυτή είναι εν μέρη και η προσιθέμενη αξία αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων σε σχέση με τι επιχορηγήσει. Γιατί οι επιχορηγήσει πολύ δύσκολα μπορεί να, να τις παρακολουθήσεις, διότι το δάνειο έχει έναν δανειστή και έναν οφειλέτη. Και ο οφηλέτης θα πρέπει να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να πείσει το δανειστή ότι θα το αποπληρώσει το δάνειο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα είδος πειθαρχίας αν θέλετε προκειμένου. Έπειτα δικασίες προσφυγής αν μπορεί κανείς να εφεσιβάλει μια απόφαση, ναι, μπορείτε να δείτε στο δικό μας website ε, λεπτομέρειες για το μηχανισμό ε, άσκησης έφεσης κατά τέτοιων αποφάσεων. Για το θέμα της ε, αξιολόγησης, του rating, είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα, περισσότερο από ποτέ σήμερα. Ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη με την αξιολόγηση τη ψηλοπτική ικανότητα των κρατών μελών και κάπου εκεί λιγάκι τα μπερδεύουμε. Ε, δηλαδή, ποιο είναι ο ρόλο των εταιριών rating, α μην το συζητήσουμε αυτό, και έπειτα η ερμηνεία αυτών των αξιολογήσεων που δίνονται σε εταιρείε και σε project. Πάντω, εν τέλει, πρέπει να αξιολογηθεί αν θέλετε η δυναμικότητα, η αποδοτικότητα ενός project, ενός δανείου. Είναι ένα δημοκρατικός τρόπος, αν θέλετε, λειτουργίας. Μπορεί να μην είναι ε, ιδανικό το σύστημα της αξιολόγησης, αλλά δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο σύστημα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτω εγώ τα θέματα που μπορώ να απαντήσω και να δώσω στον συνάδελφο να απαντήσει στα άλλα ερωτήματα για τα PPP. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο υπόλογες είναι αυτές οι υπηρεσίε οι οποίες προχωρούν σε εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. Ξεκινώντας από αυτό που έθεσε ο κύριος Γκρόλ, αν υπάρχει πράγματι ανάγκη για μια διαφορετική, για αλλαγές στον τομέα των κανόνων σε σχέση με τις δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στις αγορές, τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος μέχρι τώρα έχει εξελιχθεί αρκετά θα έλεγα όμαλα και από την άλλη αν ακούμε πραγματικά το τι λέει ο ιδιωτικός τομέας και η βιομηχανία. Αυτό που ακούγεται είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός νόμος ενιαίος για τα PPPs γιατί από ό,τι λένε το σύστημα ως έχει μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά λειτουργεί, λειτουργεί σωστά. Και οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με τις πρακτικές και σε σχέση με τους στόχους και σε σχέση με την οριμότητα των αγορών είναι επαρκώς διαφορετικές έτσι ώστε να επιτρέπουν κάποιες δυναμικές εξελίξεις και όχι να οδηγούμεθα σε ενιαίες λύσεις. Αν δει κανείς προσεκτικά αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, θα κατανοήσει ότι η εξέλιξη της χρήσης ε, των PPP στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία θα δείτε ότι έχει υπάρξει προσαρμογή σε διαφορετικά πρότυπα, κάθε αγορά έχει μάθει από την προηγούμενη και όλες οι αγορές έχουν ωφεληθεί από τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες αν θέλετε ε, ε, από τις υπόλοιπες αγορές. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης των PPP, στο έθεσε ο κύριος Ελκαντράουι. Αν κοιτάξει κανείς το σύνολο των επενδύσεων, του ύψους των επενδύσεων, θα δει κανείς ότι μπορούν να καλυφθούν και από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τους ιδιώτες επενδυτές το ότι εμείς βελτιώνουμε τη διαθεσιμότητα των επενδύσεων στη μία πλευρά της αγοράς, αυτό δεν σημαίνει ότι η άλλη πλευρά δεν πρέπει να κάνει την προσπάθειά της. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, σε κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές. Τα PPPs λοιπόν έθεσαν στη διάθεση της αγοράς κάποια χρήματα ε, κάτω από συνθήκες που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάλογα με την εθνική κάθε φορά κατάσταση, με τους κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Η ανησυχία σας ότι τα PPP σημαίνουν ότι αναλαμβάνει τους κινδύνους αποκλειστικά ο δημόσιος τομέας, αν πράγματι ε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα γιατί κάποιες εθνικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές που έχουν παίξει κάποιο ρόλο θα μπορούσαν να δεχθούν αυτού του είδους ε, την ε, κατανομή κινδύνων. Δεν είναι έτσι. Θα έλεγα ένα από τα άγνωστα κέρδη του συστήματος είναι ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές και υπάρχουν θα έλεγα αποτελέσματα τα οποία ελέγχονται επί τη βάση συγκεκριμένων αποδείξεων έτσι ώστε να καταλάβουμε και τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το συνολικό κόστος, σε σχέση με τον χρονισμό της πληρωμής, ε, ε, της κάλυψης του κόστους, αλλά και σε σχέση με την κατανομή των ευθυνών ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Η σύραγγα της μάχης, πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα PPP, αλλά δεν ήταν ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν μια απλή ιδιωτική επέμβηση. Πρέπει λοιπόν να πούμε με μια κάποια δυσκολία ότι είναι μία από τις ε, πιο ε, επιτυχείς οικονομικές επενδύσεις για το κοινό, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η επένδυση αυτή για την τραπεζική κοινότητα η οποία στήριξε το έργο. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα με λίγο διαφοροποιημένο τρόπο. Για την κυρία Μάισνα, για το αν η Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει επαρκώς την αγορά των PPPs. Εγώ θα επανέλθω στην αρχική συζήτηση. Θα πω ότι και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο κρατηδίων και σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων στη Γερμανία ακολουθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν έχουν γίνει πολλά σε σχέση με τα PPP, αλλά σε επίπεδο κρατηδίων και σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων υπάρχουν ε, υψηλά επίπεδα χρήσης των PPP σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή αυτή δεν είναι καλή ή κακή. Είναι μια επιλογή η οποία λειτουργεί σωστά για τη συνταγματική τάξη στην Γερμανία. Αντίστοιχα γίνεται και στην Ισπανία θα δείτε διαφορετική αντίληψη για την χρήση των PPP στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ότι υπάρχει λοιπόν ευελιξία, το ότι υπάρχει πλουραλισμός, αυτό γίνεται για να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές οι δημόσιες αρχές της κάθε χώρας. Νομίζω ότι συνεχώς όλες οι χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τις επιλογές τους. Για την κυρία Φώστερ και για τα JTI. Πράγματι θα συνεχίσουν τα προγράμματα αυτά. Είναι μια πολύ ειδική μορφή PPP, είναι μια συμβατική μορφή, βασίζεται στην κατανομή του κόστους και των κινδύνων και όχι στην κατανομή των εσόδων. Εδώ μιλάω σε ανθρώπους που γνωρίζουν από μεταφορές και θα ήθελα να πω ότι το κόστος χρηματοδότησης της καινοτομίας μέσω των PPP είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα είναι αναπόσπαστο τμήμα της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές πλέον. Κάθε μορφή έρευνας, κάθε μορφή βελτίωσης των υποδομών, όλες οι εξελίξεις στον τομέα της, παραγωγής της καλύτερης χρήσης της ενέργειας, της μεταφορές, όλα αυτά περνούν από τα JTI πολλές φορές και υπάρχουν πολλές γενικές διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστηρίζουν ε, την χρήση των PPP για τις καινοτομίες στον τομέα των μεταφορών. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Τέλος, Πρόεδρε, για τον κύριο Κράμα. για το αν κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια πολύ άνηση σχέση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και αν τα προγράμματα τα οποία φέρει εις πέρας ο ιδιωτικός τομέας είναι κερδοφόρα και αυτά που φέρει εις πέρας το δημόσιο είναι καταστροφικά οικονομικά. Δεν είναι έτσι, τα πράγματα αλλάζουν. Οι δημόσιες αρχές ακόμα και στις χώρες που έχουν υψηλή αξιολόγηση έχουν κάποιο όριο σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία μπορούν να δώσουν για να καλύψουν κάποιες μορφές επενδύσεων. Από την άλλη έχουμε κεφαλαιαγορές και σε ευρώ και σε άλλα νομίσματα ε, αρκετά ισχυρές. Έχουμε πολύ ισχυρές πιστοτικές αγορές. Έχουμε συνεπώς την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλούς πόρους ανάλογα με την κατανομή των κινδύνων και των ευθεριών που επιλέγουμε κάθε φορά. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει. Είδαμε ότι έχουν υπάρξει τουλάχιστον πέντε χώρες οι οποίες έχουν όριμες αγορές PPPs πλέον. Είδαμε όμως επίσης ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία και στην γειτονία μας και η Τουρκία επιταχύνουν τη συμμετοχή τους στα PPP ακριβώς γιατί θεωρούν ότι τις βοηθά τις χώρες αυτές να πετύχουν αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν όταν δεν έχουν τα PPP στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ. Έχω τέσσερις ομιλητές. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Δύο λεπτά. Μην ξεχνάτε. ότι ενώ το κοινοβούλιο λειτουργεί βεβαίω διότι όλοι έχουν το δικαίωμα να με μιλήσουν επί παντό επιστητού, αλλά παρακαλώ μην υπερκαλύπτεστε, μην επαναλαμβάνεστε. Ο κύριος Κανσιάν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτούνται κάποιες εξηγήσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το σύστημα PPP. Επιτρέψτε μου να εστιάσω τη σύντηση στο εξή σημείο. Σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 32 δισεκατομμύρια το 2020 τις μεταφορές και 50 για τις υποδομές. Συνολικά μάλλον 50 δισεκατομμύρια για τις υποδομές και 32 εξ αυτών είναι για τις ε, ε, μεταφορές. Ρωτώ λοιπόν, αν αυτά τα 32 δις μπουν σε ένα ταμείο με αυτό το σύστημα της μόχλευσης, δηλαδή με το μηχανισμό που εσείς μας περιγράφετε τι θα μπορούσαμε τελικά να καταλήξουμε να έχουμε για τις υποδομές, χωρίς τελικά να καταλήξουμε στις επιχορηγήσεις. Διότι ναι, χρειαζόμαστε το σύστημα των εγγυήσεων, όμως όταν δεν καλύπτουμε το 100% της επένδυσης, πρέπει να υπάρξει άμεση συμμετοχή ε, στη χρηματοδότηση των επιμέρους ε, προγραμμάτων δεν αρκεί, δεν αρκεί να διευκολύνουμε ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Λέω λοιπόν, άλλο το PPP που διευκολύνει, αν θέλετε, την πίστοση και κατανοώ το σύστημα του 2014 ε, που κάνετε το πιλωτικό project και Ρωτώ όμω από την άλλη, πώ θα υπάρξει άμεση συμμετοχή μέσω ενό μηχανισμού, μέσω ενό τέτοιου ταμείου που σα ανέφερε. Ποια είναι η γνώμη σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις. Καταρχάς, η δομή. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μία έξεση αξιολόγησης ε, που, μπορούν να, εξετάσουν οι επενδυτές. Υπάρχουν άλλα, άλλες εκθέσεις που αναφέρονται στην αντιστάσμιση και σε διάφορες... Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείται με ασκήσεις, αντιστάθμισης και εάν οι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα κοινά προγράμματα είναι με ιδιώτες ή μεγάλες ε, ε, ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις περισσότερο. Τρίτον, μέχρι τώρα τα PPPs ήταν εκτός ισολογισμών, το λεγόμενο off-balance όπως είπατε και ε, τώρα αυτό το στοιχείο δεν ε, ισχύει πλέον διότι στο παρελθόν όντας εκτός ε, ισολογισμών αυξάνονταν τα χρέη. Υπήρχε ο κίνδυνος αύξησης του υπερδανισμού και της υπερχρέωσης με τα ομόλογα έργων και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας πώς θα αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Η κυρία Ντουράν, δύο λεπτά. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τις ερωτήσεις των υπολείπων. Ένα μεγάλο τμήμα της εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει χρησιμοποιείται για την κατανομή του κινδύνου ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και υπάρχει και το κόστος της εμπειρογνωμοσύνης για το μοντάρισμα του προγράμματος. Αυτό επηρεάζει αρνητικά το κόστος του προγράμματος ή όχι. Δεύτερον, στα πλαίσια ποιου προγράμματος έχει υπάρξει, θα έλεγα, μια αποτυχία την οποία να αναλάβει ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτήν, την αποτυχία η τράπεζά σας. Και τρίτον, όταν μιλάτε για κριτήρια, δεν έχουμε μιλήσει για κριτήρια επιλογής. Υπάρχουν και τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι στόχοι καλύπτονται από την πολιτική εξουσία, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε. Μετά από αυτό κάνετε εσείς κάποιες αξιολογήσεις. Όταν εσείς υποστηρίζετε οικονομικά, σαν παράδειγμα, την χρηματοδότηση ενός αυτοκινητοδρόμου, λαμβάνετε υπόψη ότι στα πλαίσια αυτού του νέου αυτοκινητοδρόμου θα υπάρξει αποδυνάμωση άλλων αηφόρων, θα έλεγα, μορφών μεταφοράς προς τον αυτοκινητόδρομο και έτσι θα δημιουργηθεί ένα περιβαλλοντικό χρέος. Το λαμβάνετε υπόψη σας αυτό. Και τέλος, τέλος ο κύριος Ρίκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, δύο διευκρινήσεις μάλλον. Η πρώτη αφορά τα project bonds και η άλλη αφορά τα PPPs. Για τα project bonds. Τελικά θα υπάρξει ένας τύπος, ε, δεδομένος τύπος project bonds για κάθε πρόγραμμα ή μήπως κάθε πρόγραμμα θα δημιουργήσει αν θέλετε ειδικού τύπου project bonds. Θα υπάρξει επίσης ε, κατανομή των spread από πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των ερωτήσεων μου. Το δεύτερο κομμάτι, τα PPPs δεν λειτουργούν μόνο από τις επενδύσεις αλλά και κατά τη λειτουργία τους. Ε, έχει σημασία η διάρκεια της λειτουργίας, έχει διάρκεια η απόδοση ε, του προγράμματος και η απόσβεση του προγράμματος και των επενδύσεων. Και δεύτερον, υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς για τα PPP σε σχέση με τις επενδύσεις αυτές, δηλαδή τα χρέη τα οποία έχουν σχέση με τις επενδύσεις που εγγράφονται στην Ευρώπη, στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει κατανομή και στους δύο, να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεκρέαν, μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα απαντήσω στις ερωτήσεις που δεν συνδέονται άμεσα στα PPP. Καταρχάς ε, το στοιχείο της μόχλευσης. Πράγματι, είναι βασικός, ε, η βασική αιτία για την οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα αυτό, αυτή η μόχλευση, αυτό το εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύτιμο ανάλογα με το στοιχείο για το οποίο προορίζεται. Παραδείγματο χάρη αν είναι μετοχικό κεφάλαιο, αν είναι, ε, έργα, ε, ε, ομόλο, αν είναι ομόλογα έργων ή αν είναι ένα άλλο χρηματοοικονομικό μέσο, δεν υπάρχει πάντοτε η ίδια αύξηση του ποσοστού ή το ίδιο ποσοστό μόχλευσης, ανάλογα δηλαδή. Εσείς αναφέρω αφιερώσετε σε ένα επενδυτικό ε, ε, μέσον, σε ένα επενδυτικό ταμείο. Παραδείγματο χάρη το Margaret Fund, το οποίο είναι ε, ένα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να χρηματοδοτεί έργα υποδομών. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όμως μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται χρόνος. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται και εδραιώνεται αυτό το μέσο της μόχλευσης μέχρι του σημείου που αποφέρει αποτελέσματα χρόνος. Στο, στην άλλη ερώτηση του κυρίου Ντεμπάκε για το πώς μπορούμε να επενδύσουμε, να ε, μαζέψουμε μετρητά cash για τα ομόλογα έργων, είπα ότι αυτά τα ομόλογα είναι ήδη ο, ένας πρώτος ε, τρόπος ε, να μπορέσουμε να ε, συλλέξουμε μετρητά εκεί όπου χρειάζονται. Και η δομή την οποία χρησιμοποιούμε έχει σχεδιαστεί ακριβώς έτσι, ώστε με τους εσωτερικούς κανονισμούς να επιτρέψει στους επενδυτάς που θέλουν με μετρητά να επενδύσουν σε αυτά τα ομόλογα έργων η καινοτομία. Είναι ένα καινοτομικό αυτό προϊόν και η καινοτομία είναι σημαντική όχι μόνο στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντική στον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτομικές πτυχές των μεταφορών. Αυτό λοιπόν ε, το μοντέλο επικεντρώνεται ακριβώς σε, σε στις μεταφορικές δυνατότητες χρησιμοποίησης. Ε, στην επόμενη ερώτηση, το κόστος της εμπειρογνωμοσύνης, της προετοιμασίας της, στα περισσότερα ε, ε, έργα, αυτό το κόστος έχει συνυπολογιστεί στο γενικό κόστος. Μόνο στο, στο πρόγραμμα Jaspers, Υπάρχει μία εξαίρεση διότι το Jaspers ε, σχεδιάστηκε από την αρχή ως δωρεάν υπηρεσία για να προετοιμάσει ε, κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους ε, να διαμορφώσουν τέτοια προγράμματα. Αλλά σε όλα τα άλλα γενικά έργα συνυπολογίζονται αυτό το κόστος προετοιμασίας και σχεδιασμού. Η κυρία Ντυρό επίσης αναφέρθηκε σε περιβαλλοντικά κριτήρια. Σας διαβεβαιώ ότι τα περιβαλλοντικά κριτήρια είναι εξαιρετικά σημαντικά, τα λαμβάνουμε υπόψη και έχουμε ολοκληρώσει μαζί με το Κοινοβούλιο μία ευρύτατη ε, διαβούλευση για να καθορίσουμε ποια είναι τα καλύτερα κριτήρια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ε, για τα έργα μας, για την αξιολόγηση των έργων μας και όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Γιατί ξέρετε, το περιβάλλον δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι απόλυτα διαφανής αυτή η προσέγγιση μας στα περιβαλλοντικά κριτήρια και θέλω να τονίσω και μετά από αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε διότι και ο πρόεδρος μας το υποστηρίζει αυτό πλήρως, η τράπεζα θέλει να, είναι, ε, ε, να χειρίζεται όλα τις τα θέματα με απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη ευθύνη, να είναι υπόλογος ε, δηλαδή στο ελεγκτικό συνέδριο, στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ας τονίσω και κάτι άλλο. Το διοικητικό μας συμβούλιο που εγκρίνει με μονομένο έργο έχει 28 μέλη, ένα από κάθε κράτη μέλος και ένα από την Κομισιόν. Και εξετάζουμε έργα μόνο ε, μετά από την φάση αξιολόγησης των εσωτερικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει και την Κομισιόν. Γι' αυτό ακριβώς, αφού έχει γίνει ο ενδελεχής έλεγχος ε, των αιτήσεων και έχουν εγκριθεί τα έργα αυτά, εν συνεχεία πηγαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και το ξαναεξετάζουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος ε, Μπάνετ. Ε, αφορά τώρα τη χρησιμοποίηση αυτού του μέσου είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τις δομές του PPP με μεγάλη επιτυχία για να συγκεράσουμε τα δημόσια και τα ιδιωτικά διαθέσιμα κεφάλαια. Και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Απαντώ στον κύριο Ντεμπάκα για το, τα υπέρ και τα κατά του εντός ή εκτός ισολογισμών, on-off balance. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι εάν οι άνθρωποι βασιστούν απόλυτα για τα κριτήρια αξιολόγηση στο on ή off ε, balance, δηλαδή sheet, στο εντός ή εκτός ισολογισμό, κάνουν λάθος προσέγγιση για, για να κρίνουν τα PPP δεν πρέπει αυτό το στοιχείο, αν είναι εντός ή εκτός προϋπολογισμού, να είναι το κρίσιμο στοιχείο και το απόλυτο για την αξιολόγηση. Το θέμα είναι τα χρέη πρέπει ε, να αναγνωρίζονται, να είναι καταγεγραμμένα σε κάποιο χαρτί, σε κάποιον ισολογισμό, ή στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο μέρος του έργου. Άρα, λοιπόν, ε, αναγνωρίσουμε ότι κάπου πρέπει να είναι καταγεγραμμένα τα, ε, τα δάνεια, τα χρέη. Ε, αλλά αν είναι γραμμένα εντός ή εκτός ισολογισμού δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για την απόφαση. Κυρία Ντιμό, δεν, δεν υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος αποτυχιών, μακρύς κατάλογος και είμαστε, θα έλεγα, ε, ίσως θα έλεγε κάποιος ότι είναι λίγο απογοητευτικό που δεν έχουμε ένα μακρύ κατάλογο λαθών και σφαλμάτων. Έχουμε ε, διαπιστώσει, έχουμε ε, πολλές επιτυχίες, έχουμε εφαρμόσει με επιτυχία πολλά προγράμματα και έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία αξιόπιστα. Τώρα, υπάρχουν πολλοί ιδιώτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πετύχουν το μέγεθος των αποδόσεων που ήλπιζαν. Ε, και υπάρχουν επίσης πολλοί δημόσιοι τομείς που ξεπέρασαν τους προπολογισμού τους. Η... Εάν τώρα ένα έργο είναι ε, θετικό ή αρνητικό, αυτό κρίνεται από τη σύμβολή του στο δημόσιο τομέα και στο τι όφελος έχει πετύχει ως προς τους γενικούς στόχους του. Αλλά μετά αυτά που ο Κράμερ για το, τη σύραγγα της μάχης, ε, αυτό ήταν ένα παράδειγμα όπου οι προσδοκίες του κοινού ήταν α και οι χρηματοοικονομικές προσδοκίες ήταν β, τελείως διαφορετικά. Αλλά εάν ρωτήσετε τους χρήστες της σύραγγας της μάχης για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις καλυτέρευσε σημαντικότατα ε, τις ροές ε, των επιβατών και των μεταφορών μεταξύ των του Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ήταν λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θετικό αποτέλεσμα αυτό, παρόλα τα χρήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα που είχαμε. Το, τελικό όφελος ήταν θετικό. Γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, δεν έχουμε έναν μακρύ κατάλογο ε, μεγάλων αποτυχιών, θεαματικών αποτυχιών. Ευχαριστώ η συνθήκη του Canterbury του μεσαίωνα δηλαδή. Είναι ακριβώς το πρόβλημα που είχαμε πάντοτε με το μπλοκάρισμα της επικοινωνίας μας μέσω της σύραγγας. Λοιπόν, η συνθήκη του Κάντερμπορι αυτή είναι που μας παρουσίασε τα προσκόμματα. Μέχρι τώρα, ε, παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει γερμανικό τρένο που περνάει τη σύραγγα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα μέλη στα θέματα τα οικονομικά, τα θέματα των χρημάτων. Υπάρχει μεγάλη δυσπιστία από πλευράς των ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρχών σε αυτά τα προγράμματα. Όμως εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλες αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και τον καιρό που διαθέσατε.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στη μέρη διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με μελέτη σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε θαλάσσιους λιμένες. Ζήτησε η Επιτροπή μας πέρυσι αυτή τη μελέτη ώστε να δούμε κατά πόσον οι φυστάμενοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων ε, ισχύουν και εφαρμόζονται ε, πλήρως και στα θέματα των θαλάσσιων λιμένων ή χρειάζονται καθευτήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις εν προκειμένου. Ο κύριος Βαν Ρόι έκανε τη μελέτη, ο οποίος πολύ ευγενικά ήρθε εδώ δίπλα μου. Παρακαλώ, 15 λεπτά σας δίνω να μας παρουσιάσετε αυτή τη μελέτη. Και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα θέσουν ερωτήσεις. Ξέρετε, να μιλούμε για τις θαλάσσιμες μεταφορές λίγο πριν τα Χριστούγεννα είναι αρκετά δύσκολο και βαρύ θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Βανρόη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις στα αγγλικά, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω την παρουσίαση στα Ολλανδικά, καθώς είναι η μητρική μου γλώσσα. Κύριε και κύριοι, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα, για την παρουσίαση των ευρημάτων αυτής της μελέτης στην Επιτροπή σας. Είναι μία ευσύνοπτη μελέτη για τις κρατικές ενισχύσεις για τους θαλάσσιους λιμένες. Ελπίζω... υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο μου, οπότε θα πρέπει να πάω λιγάκι πιο δεξιά και να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο του Προέδρου. Δύο θέματα θέλω να επισημάνω. Πρώτα απ' όλα είναι ότι οι κρατικές συνεχίσεις είναι ένα θέμα ευρύτατο και θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο διάγραμμα. Λοιπόν, όπως μόλις είπα, οι κρατικές ενισχύσεις είναι κάτι ευρύτατο, καλύπτουν μια πλειάδα υπηρεσιών και υποδομών. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας στις κρατικές ενισχύσεις για τις υποδομές που αφορούν τους θαλάσσιους λιμένες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μέθοδο ανάλυση που χρησιμοποιήσαμε. Το δεύτερο που αναρωτηθήκαμε ήταν το εξή. Πώς μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα την ε, ανταγωνιστική θέση των λιμένων ε, της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης. Δηλαδή, οι κρατικές ενισχύσεις επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των λιμένων στον Βορρά και τον Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις αυτή τη στιγμή υιοθετήθηκαν με τη μορφή που έχουν πάνω κάτω σήμερα τη δεκαετία του 1990 και θυμάμαι ε, τον προκάτοχο της ΓΔ Move που είχε κάνει την πρώτη πρόταση του 1992 και μετά είχαμε μία σειρά διαδοχικές εκθέσεις ε, για αυτό το ζήτημα γιατί το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα κρατικών ενισχύσεων και ε, η αλήθεια είναι ότι έω σήμερα δεν υπήρξε μία σημαντική πρωτοβουλία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τους θαλάσσιους λιμένες. Φαίνεται λοιπόν ένα θέμα που δεν έχει απασχολήσει, δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα ακόμη, όμως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων την ανταγωνιστικότητα και των επιχειρήσεων. Αναγκαστικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να σας δώσω το γενικότερο πλαίσιο σχετικά με κάποια ναυτιλιακά στοιχεία και τους θαλάσσιους λιμένες, γιατί είναι καλό να έχουμε μια γενικότερη εικόνα και μετά θα περάσω στα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Λοιπόν, αν δείτε αυτό το διάγραμμα, βλέπετε τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή πώς έχουμε την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και τα διαφορετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΑΕΠ. Βλέπετε την τελευταία δεκαετία μία φοβερή επιτάχυνση λόγω της παγκοσμιοποίησης με αποτέλεσμα να αυξηθεί, αν θέλετε, πολύ η ζήτηση για, το, για καλύτερο και μεγαλύτερο δυναμικό στις υποδομές των θαλάσσιων λιμένων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ζήτηση για μεγαλύτερο δυναμικό, οπότε αναγκάζονται ε, τα λιμάνια, λόγω της παγκοσμιοποίησης, να ανταποκριθούν σε αυτή την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Πώς όμως όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε ένα πεδίο ίσων ευκαιριών, με θεμητούς όρους για όλους, χωρίς να υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Άρα, θα πρέπει οι χρηματοδότες των υποδομών να γίνουν με την απόλυτη τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Θα δείτε όμως την προσοχή μου ότι τελικά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό πλήρως. Βλέπετε τώρα σε αυτή τη διαφάνεια τη συνέπειε, τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στους διάφορους τομείς των ε, φορτίων, των κάργο που παίρνουν τα λιμάνια μας. Και βλέπετε ακριβώς ποιος είναι ο κύριος όγκος εργασίας στα θαλάσσια λιμάνια και βλέπετε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη προσβασιμότητα για το εμπόριο με εμπορευματοκιβώτια στα θαλάσσια λιμάνια. Δημιουργείται λοιπόν συνήθως μια πολύ περίπλοκη κατασκευή ε, στους θαλάσσιους λιμένες για να εξυπηρετηθούν διάφορες μορφές εμπειρίου, αλλά όταν μιλάμε μόνο για τα κοντέινερ, για τα εμπορευματοκιβώτια, οι υποδομέ που απαιτούνται είναι διαφορετικέ. Γιατί συνήθω ε, με τα εμπορευματοκιβώτια χρειαζόμαστε τι συνδυασμένε μεταφορέ και εκεί δεν τίθεται μόνο το θέμα τη υποδομή, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πολύ εξειδικευμένη ζήτηση για ε, συγκεκριμένες υποδομές στους θερματικούς σταθμούς των λιμένων για την υποδοχή των κοντέινερ. Αυτό σημαίνει, συνεπάγεται, πολύ μεγάλες ε, επενδύσεις για να μπορέσει να αγκυροβολήσει ένα μεγάλο πλοίο ε, με εμπορευματοκιβώτια χρειάζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, πολύ δαπανηρές. Και βεβαίω, ε, για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλοι, τεράστιοι όμιλοι που επενδύουν ακριβώ σε αυτόν τον τομέα. Στην κατασκευή των κατάλληλων υποδομών για τα κοντέινερ. Βεβαίω, ο παράγοντας της ε, οικονομικής μη προβλεψιμότητα είναι πολύ σημαντικός εν προκειμένου. Και Γι' αυτό απαιτείται από τον επιχειρηματικό κόσμο όλοι εμείς να έχουμε απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων προκειμένου. Έπειτα μίλησα πριν για την... τον ανταγωνισμό και τις διαφορές όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των λιμένων στη Βόρεια και την Νότια Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μια γενική εικόνα της κατάστασης των εξειδικευμένων υπηρεσιών στα λιμάνια. Βλέπετε εδώ τη βόρειο διάσταση και την Μεσόγειο από την άλλη πλευρά. Βλέπετε ότι τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες λιμένων που τις σκεγγραφούμε με πορτοκαλί και πράσινη γραμμή. Βλέπετε την ένταση των, ε, της κινητικότητας στην ε, Βόρεια Ευρώπη που είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι συμβαίνει στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπουμε αυτή τη διαφορά στην κινητικότητα, γιατί είναι διαφορετικά πρώτα απ' όλα ε, τα είδη των σκαφών που πλέουν στις περιοχές αυτές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ιστορικούς λόγους. Ιστορικός πώς οι βόρειοι λιμένες είναι πιο κοντά σε βάσεις διοικητικής επιμελητίας σε σχέση με τα λιμάνια του Νότου. Η Κίνα, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο λογικό να γυροβολήσει στο Τζόια Τάουρο ή στη Γένοβα ή στη Μασαλία. Και μετά να μεταφορτωθούν τα κοντέιρερ και να πάνε ο σου στη Βόρεια Ευρώπη αν κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς, ένα μεγάλο ε, σκάφος μπορεί να μεταφέρει έως και 15.000 κοντέινερ. Ενώ ένα τρένο μπορεί να μεταφέρει μόλις 80 ε, Άρα κατανοείται τη συμφόρηση στις οδικές και δρομικές μεταφορές για να μπορέσουν να μεταφερθούν οδικός ή δρομικός όλα αυτά τα κοντέινερ από την Νότια στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα η προτιμόμενη λύση είναι να πάνε κατευθείαν τα σκάφη στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. τελικά είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι να εκφορτώσουν στα λιμάνια της Ότας Ευρώπης και να μεταφερθούν τα εμπορεύματα συνδρομικά και οδικά. Έπειτα, η εμβέλεια της διασύνδεσης που έχουν τα λιμάνια με την ενδοχώρα. Η, η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει πολύ ε, εδώ και για μεγάλο διάστημα. Βλέπετε βεβαίως ότι υπάρχει και ένα μέσος χώρος, μια μέσα ζώνη όπου υπάρχει επικάλυψη της εμβέλειας ε, της διασύνδεσης των λιμένων. Είναι, αν θέλετε, σαν ε, αμφισβητούμενες ε, ή μάλλον είναι οι ζώνες που τις, θέλουν να τις κατακτήσουν όλοι. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη που βλέπετε στην κεντρική Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ένα ε, συντηρητικό πλεονέκτημα, αλλά τελικά είναι πολύ περιορισμένης εμβέλειας. Αν το δούμε όμως με τη φωνή της λογικής, υπό όρους. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά εν προκειμένου ώστε να λειτουργήσει προς όφελος, αν θέλετε, των λιμένων του Βορρά ή του Νότου. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για ανταγωνισμό ανάμεσα στα λιμάνια του Βορρά και του Νότου, αλλά ανάμεσα στα λιμάνια του ίδιου βελληνικού ίδιας εμβέλειας, αν θέλετε, ανάμεσα στο Ρότερταμ και την Αμβέρσα ή ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Μασαλία. Εκεί ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο σκληρός. Άρα ο ανταγωνισμός στο λιμένο στην ίδια Λεκάν είναι πολύ πιο ισχυρός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των γειτόνων είναι πολύ πιο έντονος. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζω εγώ ως λιμένας τους κανόνες του παιχνιδιού για να ξέρω πώς θα αγωνιστώ ε, εντός ενός θεμητού πλαισίου ε, τους γειτονικούς λιμένες και πώς θα επενδύσω ε, στις λιμενικές υποδομές χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες κρατικών ισχύσεων. Και πάω στην επόμενη διαφάνεια στα συμπεράσματα. Μίλησαμε για, την, για τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα, την προσβασιμότητα των, ε, του εμπορίου και λόγω τη παγκοσμιοποίηση, την αυξανόμενη συνεχώ ζήτηση σε μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά τι υποδομές στα λιμάνια και να βγει όλο αυτό απαιτείται μεγάλη διαφάνεια και ίση όρη ε, ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων. Τώρα να περάσω στο δεύτερο τμήμα. Τις ίδιες κρατικές ενισχύσεις. Ε, Εδώ βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια project που ξεκίνησαν το 2009 σχετικά με το δυναμικό των λιμένων για την υποδοχή εμπορευμα... εμπορευματοκιβωτίων. Στην παρουσίαση αυτή μιλώ συνεχώς για τα κοντέινερ, για τα εμπορευματοκιβώτια. Όμως ε, οι λιμένες περιέχουν ε, μια σειρά υποδομών που δεν αφορά μόνο τα κοντέινερ. Χρειάζονται υποδομές κατάλληλες για την ε, αγκυροβόληση των σκαφών, ε, τους ε, λιμενοβραχίονες, την υποβοήθηση της πρόσβασης μεγάλων φορτηγών για τη διασύνδεση με τις οδικές μεταφορές, άρα υποδομές για την εκφόρτωση, μεταφόρτωση φορτίων Επίσης υπάρχουν και υπερκατασκευές ε, στους λιμένες όπως είναι η γερανή και πώς εξοπλισμός. Οι υπερκατασκευές λοιπόν που είναι η γερανή και όλοι οι μηχανισμοί για την εκφόρτωση-μεταφόρτωση είναι ένα εξίσου μεγάλο κομμάτι όταν μιλούμε για υποδομές ε, στους λιμένες. Οι κρατικές ενισχύσεις λοιπόν αφορούν όλες αυτές τις κατηγορίες υποδομών και για τις υπερκατασκευές και για τις υποδομές όπως και για τις πολλαπλές ε, ή χωριστές χρήσεις ε, των λιμένων. Στην επόμενη διαφάνεια. Οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι νομικός, Είμαι οικονομολόγο. Σω θα πρέπει να έχω και νομικέ γνώσεις. Οπότε δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα νομικά ερωτήματα, ούτε μπορώ εγώ να δώσω ένα νομικό ορισμό των κριτικών ισχύσεων. Υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα. Όμω, το, το άρθρο 107 της ε, συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση, το παλαιό άρθρο 87 τη συνθήκη. ε, ε, ρυθμίζει τα τοπικών ισχύσεων. Το άρθρο 107 αποτελείται από τρει παραγράφου και εκεί ορίζονται οι μη συμβατέ κρατικέ ενισχύσει. Και η παράγραφος 1 μιλάει για τη μεταφορά δημόσιων κονδυλίων που λειτουργεί επωφελία μίας επιχείρησης Επίσης, οι κρατικές ενισχύσεις λειτουργούν επιλεκτικά, άρα κάνουν, μία, κάνουν διακρίσεις και άρα οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και η στρέβλωση του ανταγωνισμού έχει συγκεκριμένε συνέπειε για του εμπόρου. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια που πρέπει να λειτουργήσουν σωρευτικά θα πρέπει να υπάρχουν για να θεωρηθούν μη συμβατέ κριτικέ ενισχύσει. Το άρθρο λοιπόν 107 της συνθήκης ουσιαστικά απευθύνεται μόνο στα κράτη-μέλη και όχι στον ευρύτερο κόσμο. Άρα και ποιες είναι οι συνέπειες. Εδώ θα το είναι ερωτηματικό. Στα επόμενες παραγράφους του άρθρου 107 είναι οι de jure παρεκκλήσεις, δηλαδή σε περίπτωση θεομηνιών μπορούν να προβλεθούν οι κρατικές ενισχύσεις όπως και άλλες παρεκκλήσεις ε, διακριτικού χαρακτήρα που προβλέπονται από το άρθρο 107. Παρεκκλήσεις μπορούν να υπάρξουν για διάφορους λόγους όταν έχουμε να κάνουμε με ένα έργο ευρύτερης κοινή ωφέλεια ή αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας που χρήζει ενίσχυσης, ενδυνάμωσης τέτοιου είδους ε, είναι οι παρεκκλήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 107 σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ότι στην παράγραφο 1 ποιες είναι οι μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και οι παράγραφοι 2 και 3 της παρεκκλήσεις. Το πρόβλημα όμως πολύ συχνά είναι στην πράξη ότι όλοι επικαλούνται στις παραγράφους 2 και 3 όταν θα πρέπει να περάσουν από τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο έχουν τηρηθεί κανόνε κρατικών ισχύσεων. Όλοι επικαλούνται λοιπόν τι παρεκκλήσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 107. Και αν δεν υπάρχει και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πολύ συχνά αναπαράγεται αυτό το κακό ε, μοντέλο. Υπάρχει λοιπόν μια παρερμηνία, αν θέλετε, ε, από πολλές ε, πλευρές σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών τι κάναμε. Επιλέξαμε εννέα χώρες και τα θαλάσσια λιμάνια τους για να κάνουμε αυτή τη μελέτη. Η επιλογή αυτών των χωρών και των λιμένων ε, οφείλεται στη γεωγραφική θέση των χωρών και στις διαφορετικές κατηγορίες των λιμένων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε εδώ τις κατηγορίες των λιμένων. Είναι σημαντικό να δούμε δηλαδή, και την οργάνωση, τη διάρθρωση των λιμένων. Και επίση εξετάσαμε και συγκεκριμένε περιπτώσει κρατικών ενισχύσεων και προσπαθούμε να κάνουμε γενικότερε προβολέ. Το συζητήσαμε με διάφορους αρμόδιους πολιτικής αλλά και με τον κλάδο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε συμπεράσματα και συστάσεις που θα παρουσιάσω σε λίγο. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω λίγα λόγια για την διάθεση και την οργάνωση των λιμένων στην Ευρώπη. Να πω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα εξετάζει γενικά την οργάνωση των λιμένων και κατέληξε σε τέσσερις κατηγορίες, τέσσερα είδη λιμένων. Η πρώτη κατηγορία είναι τα δημόσια λιμάνια, τα λιμάνια που ανήκουν αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις δεν γνωρίζω αν μπορεί κανείς να ταυτίσει νομικά τις κρατικές ενισχύσεις με αυτή την κατηγορία λιμένων. Πάντως, εδώ πραγματικά θα πρέπει να είστε πολύ αυστηροί και πολύ προσεκτικοί σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Και μετά βλέπετε τις υπόλοιπες ε, κατηγορίες λιμένων που οι υποδομές στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μένουν στο δημόσιο, αλλά ε, μετά εμπλέκεται και ο ιδιωτικός τομέας. Βλέπετε λοιπόν στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία, όπου ε, υπάρχει η συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λιμανιών, το 58%, είναι η τρίτη κατηγορία, αυτά landlord ports ε, που ε, ανοίγουν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Δηλαδή σημαίνει ότι η λιμενική αρχή, εν προκειμένου σε αυτή τη τρίτη κατηγορία, είναι υπό την αιγίδα κάποιας δημόσιας αρχής, εθνικής περιφερειακής αρχής, αλλά υπάρχει ένας ιδιοκτήτης της όλης ζώνης του λιμανιού και είναι υπεύθυνο ιδιοκτήτης για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το λιμένα. Οι κρατικέ ενισχύσει που δεν συνάδουν με την εσωτερική αγορά είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο σε αυτή την κατηγορία. Στην τελευταία κατηγορία είναι τα πλήρω ε, ιδιωτικοποιημένα ε, λιμάνια, περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει ε, που είναι 0% τα δημόσια λιμάνια. Αυτά ουσιαστικά είναι ε, τα τέσσερα είδη. Αυτή είναι και η δουλειά που κάναμε. Να δούμε τώρα ποια είναι τα συμπεράσματα. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, δεν χρειάζεται αυτή, κατευθείαν στα συμπεράσματα. Μετά από συζητήσεις που κάνουμε με τους ενδιαφερόμενους του τομέα και με αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική ήταν σαφές ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να επεξεργαστούμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Το ταχύτερο θα κάνουμε σύντομα ορισμένε ανακοινώσει, αλλά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της έλλειψης διαφάνειας και της ισότιμη μεταχείρισης, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, χωρίς ε, να θέλω να είμαι υπερβολικά επικριτικός, αλλά υπάρχουν ορισμένες... Ε, προτάσεις που δείχνουν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις κρατικές ε, ενισχύσεις. Αλλά υπάρχουν πολλά προσκόμματα με, ενδοτομεακές, ε, ε, με ενδοτομεακούς ανταγωνισμούς και διαμάχες. Παραδείγματος χάρη η DG Move μέχρι το 2010 δεν υπεύθυνε για τις κρατικές ενισχύσεις για τα λιμάνια. Αυτό εν συνεχεία μεταφέρθηκε στην DG Εμπορίου, στην DG.com αυτή τη στιγμή η Γενική Διεύθυνση COM, DGCOM, κάνει μία μελέτη η οποία θα εξετάσει σε βάθος αυτό το θέμα και επί τη βάση αυτής της μελέτης θα ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία. Επίσης, ε, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι έχουμε ενισχύσει, έχουμε δείξει μια προτιμησιακή ε, συμπεριφορά έναντι των ε, λιμανιών στο Νότο, ότι έχουμε προτιμήσει τα λιμάνια στο Νότο με κρατικές ενισχύσεις. Λοιπόν, προτιμησιακή μεταχείριση καλύτερη, περισσότερες δηλαδή κρατικές ενισχύσεις για την υποδομή, για την οργάνωση κλπ. από ότι τα λιμάνια του Νότου. Όταν όμως εξετάσαμε τα ποσά και τα αριθμητικά στοιχεία των ενισχύσεων που δώσαμε, δεν διαπιστώσαμε μια τέτοια προτιμησιακή μεταχείριση ή τέτοιες διαφορές που να οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Εγώ ο ίδιος έκανα μία μελέτη και δεν διαπίστωσαν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές μεταχύσεις μεταξύ Βορρά και Νότου. Τώρα, επειδή ο τομέας αυτός είναι πολύ διαφοροποιημένος, υπάρχει από οικονομικής απόψεως προστιθέμενη ε, αξία και είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε σκληρή, τη λεγόμενη σκληρή νομοθεσία. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Επίσης, δεδομένου ότι μίλησα για τους διαφορετικούς τύπους υποδομών, η Κομισιόν έχει αναλάβει, έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να ορίσει τους τύπους των υποδομών, τις μορφές των υποδημών και τις κρατικές ενισχύσεις για κάθε κατηγορία δεν θα μπορέσετε εσείς να λύσετε το πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από μια συγκεκριμένη περίπτωση αναθεώρησης ε, του λιμανιού του Βέντσπιλς. Και εάν υπάρχει μία προβλήτα, ας πούμε, η προβλήτα, αν χτίσεις μία προβλήτα, αυτή δεν δεν προσφέρει τίποτα δεν προσφέρει τίποτα στην ε, αύξηση της εμπορικής αξίας φόρτωσης και εκφόρτωσης του λιμανιού. Όμως έχει μία αξία για άλλες λειτουργίες του λιμανιού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να ορίσουμε και να αξιολογήσουμε ένα συγκεκριμένο έργο. Τώρα, Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Πέντε συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μιλητής αλλάζει από τα αγγλικά στα ολλανδικά. Θα αλλάξω τώρα γλώσσα, λέει πάλι. Ωραία, λοιπόν. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες του τομέα για να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να διαμορφώσουμε τις κρατικές ενισχύσεις και όλα, και όλα τα συναφή θέματα για τα λιμάνια. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία με την Κομισιόν για κοινέ κατευθυντήριες γραμμές και θα συστήσουμε στο Κοινοβούλιο να εξετάσει την πολιτική ε, την πολιτική παροχών προς ε, τους φορείς που ε, λειτουργούν τους λιμένες, δηλαδή τους, ε, τους λιμενικούς οργανισμούς και τι είδους συμφωνίες μπορούν να γίνουν και ποιες είναι οι παραχωρήσεις και οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας. Πο, πολλά λιμάνια, ιδίως αυτά που είναι κάτω από 40 εκατομμύρια δεν έχουν την υποχρέωση να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για τα κονδύλια που προέρχονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό φορέα. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα διαφάνειας εδώ. Το άρθρο 117 αναφέρεται μόνο σε κράτη-μέλη και όχι σε τρίτες χώρες. Όμως για την Βόρειο Θάλασσα και ε, και τη Μαύρη Θάλασσα ε, ισχύουν διαφορετικέ ε, διατάξει διότι εκεί συνεργαζόμαστε με τρίτε χώρες. Τέλο σα ανέφερα το λιμάνι του Βέντσπιλς με την προβλήτα και τον, τη, τη δυσκολία ορισμού. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αν τα μελετήσουμε θα είναι πολύ χρήσιμα. Διάφορα, διάφορες άλλες εντυπωσιακέ λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ακριβώς ε, ποιες είναι οι δημόσιες επενδύσεις και πώς πρέπει να αξιολογηθούν από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ, ο κύριος Κράμερ, ο κύριος Ελκαντρούι. Μην ξεχνάτε, είμαστε υποχρονική πίεση. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση την οποία κάνατε. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια μικρή κριτική. Διάβασα τη μελέτη σας με μεγάλη ταχύτητα, πρόχειρα λίγο και καλό θα είναι να ελέγξει θα έλεγα τα στοιχεία τα οποία δίνεται κάποιος που γνωρίζει καλά τη Μαύρη Θάλασσα. Ίσως μερικές φορές να υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τους ορισμούς που χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στις λιμενικές υποδομές. Κάποιες από τις υποδομές αυτές έχουν ολοκληρωθεί, κάποιες άλλες έχουν υποστηριχθεί από τον δημόσιο τομέα, κάποιες όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να προσέξουμε λίγο στους όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι τα συμπεράσματα. Λέτε ότι έχουν ακολουθηθεί εντελώς διαφορετικές μέχρι τώρα πρακτικές σε σχέση με τις επενδύσεις, με τις δημόσιες βοήθειες για τη διαχείριση των λιμένων και ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες τρευλώσεις στον ανταγωνισμό. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Δεν χρειάζεται να προτείνουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Κάποιες ερωτήσεις τώρα. Αναφερθήκατε στις γενικές αρχές, αλλά από την άλλη εσείς ο ίδιος λέτε ότι κάθε λιμένας είναι διαφορετικός του άλλου. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται να γίνουν εργασίες εκβάθυνσης του πυθμένα μερικές φορές αυτό γίνεται και σε ανοιχτή θάλασσα, στους δρόμους προς τον συγκεκριμένο λιμένα. Είχα πάει και μια επίσκεψη με την Επιτροπή στη Βόρειο Αφρική και είδαμε τις διαφορές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται είναι κάποιες τρίτες χώρες να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό ε, χώρο ε, μεταφορών. Τότε θα υιοθετήσουν και τους κανόνες. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσουμε 12.30. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρούμε. Αν θέλετε να μας λέτε ιστορίες, μπορείτε. Εμείς θα τελειώσουμε 12.30. Είτε έχετε τελειώσει, είτε δεν έχετε τελειώσει. Κυρία Μάιστα. Εγώ θα είμαι πιο σύντομη. Καταρχά δεν αναφέρεται ένα λιμάνι στην, ε, στον Ιντερζάξεν, στην ε, Σαξονία που κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκά λεφτά. Εν συνεχεία υπάρχει μια περιφερειακή διαφοροποίηση μεταξύ βορρά και νότου, αλλά δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές, εγώ προέρχομαι τη Βόρεια Γερμανία και λέω ο καθένας μπορεί να διαλέξει κάτι. Στο λιμάνι του Wilhelmshaven μπορούν να έρθουν μεγαλύτεροι, μεγαλύτερα λιμάνια διότι είναι πιο βαθύ και είναι ανοιχτή θάλασσα, άλλα λιμάνια είναι πιο μικρά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν λιμάνια για τον καθένα, για κάθε ανάγκη. Δεν πιστεύω ότι οι κρατικές ε, ε, ενισχύσεις πιστεύουν περισσότερο στο νότο ίσα ίσα αντίθετα επειδή οι θαλάσσιες μεταφορές ε, το κόστος μειώνεται πιστεύω ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι πιο χρήσιμες στο βορρά θα κατευθυνθούν ισότιμα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επενδύσεις στα, στα λιμάνια, πρέπει οπωσδήποτε να το βοηθήσουμε. Και το θέμα είναι ε, εάν μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη ακόμα πιο ανταγωνιστική. Ο κύριος Κράμερ, κοιτάξτε, άμα ακούμε μία διάλεξη τριών τετάρτων, πρέπει να δώσετε περισσότερο χρόνο μιλία στα μέλη. Στη Γερμανία δεν υπάρχει μία εθνική πολιτική ε, ε, λιμένων. Ε, είναι πέντε συναρμόδια υπουργεία. Το Υπουργείο για τα Τελωνία, το Υπουργείο για το Λιμενικό Σώμα, το Υπουργείο για τα Οικονομικά, το Υπουργείο του Κρατηδίου, το Υπουργείο για την Αλία, τα Υφυπουργεία και οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες των κρατηδίων. Αυτή τη στιγμή το, το Αμβούργο παραδείγματο χάρη, το οποίο είναι μεμονωμένο κρατήδιο, θέλει να κάνει εκβάσινση του ποταμού Έλβα, αλλά δεν έχει τα απαραίτητα κονδύλια, ενώ άλλα λιμάνια παίρνουν κρατικές ενισχύσεις. Ο Παύλο Κώστα ήταν εδώ, ο οποίος διαχειριζόταν το λιμάνι στην Βενετία και οι Ιταλοί έχουν συνεργαστεί ε, η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία και είπαν ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι συνεργασία μεταξύ των λιμανιών και πρωτοβουλίες διακρατικές για να μπορέσουν να ενεργήσουν ταχύτερα. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε, έχουμε το βλέμμα συνέχεια στραμμένο προς το εξωτερικό και δεν κοιτάμε τι γίνεται μέσα στα χωράφια μας, ε, στα λιμάνια μας. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω με την τελευταία ερώτηση για τη συνεργασία, την ενδολιμενική συνεργασία. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας, ε, διότι τα λιμάνια έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το λιμάνι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος ε, πρέπει να φροντίσει τα μέλη του. Εάν λοιπόν υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός σε ένα κράτος μέλος, δηλαδή κεντρικοποιήσουμε όλη αυτή τη διαχείριση, θα πρέπει να ε, δραστηριοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε και πάρα πολλά πλοκάμια τα οποία να φτάνουν στα διάφορα άκρα. Άρα λοιπόν κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη λιμενική πολιτική και αυτή δεν υπάρχει σε όλες μας κυβερνήσεις. Πρέπει να υποχρεώσει λιμάνια να συνεργαστούν. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση. Μπορεί στο επίπεδο των λιμενικών αρχών, του λιμενικού, του management. Όμως δεν τους αρέσει να το ακούνε αυτό, διότι κάθε κυβέρνηση θέλει να κάνει τα δικά της και δεν είναι πολύ πρόθυμη να συνεργαστεί και να παραχωρήσει εξουσία. Όμως πρέπει να συνεργαστεί το Αμβούργο με τη Βρέμη, η Βρέμη ε, με το Ρότερνταμ, η Αντβέρπη με ε, το... με την Προύζ. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν αυτά τα λιμάνια, έστω και αν είναι σε άλλες χώρες, δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμένα δημόσια κονδύλια για τις επενδύσεις. Ξέρουμε όλοι ότι είναι περιορισμένες οι επενδύσεις, οι πιστώσεις είναι περιορισμένες, οι επενδύσεις στα λιμάνια μειώνονται σημαντικά και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Εάν δεν λειτουργήσουμε σε ένα υπερ εθνικό επίπεδο και αν δεν επικεντρώσουμε την πολιτική μας σε συγκεκριμένους στόχους δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Ξέρω ότι ορισμένοι εκπρόσωποι του τομέα είναι εδώ και δεν θέλουν να τα ακούν αυτά, δεν τους αρέσει. Όμως εγώ πιστεύω κάνοντα ότι η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Δεύτερον, αυτά που είπε ο κύριος Ελ Καντράουι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να εξετάσουμε τον ευρωπαϊκό τομέα, τον ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Διότι έχετε δίκιο. Αν πάμε προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα χρειαστούμε 10 χρόνια και. Άρα λοιπόν καλύτερα να διαμορφώσουμε και να στοχεύσουμε στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Περνάμε τώρα στον Αντιπρόεδρο Κάλλας. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας, γιατί όπως είπα στις 12.30 θα τελειώσουμε. Μάικολ, έχει δίκιο ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια καλύτερη δομή όταν μας παρουσιάζουν τέτοιες μελέτες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι πανεπιστημιακοί μπορεί να μας μιλάνε ώρες ολόκληρες, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που έχουμε εμείς. Εδώ δώσαμε 15 λεπτά στη διάθεση του ομιλητή και είδατε που καταλήξαμε και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έδωσα το λόγο και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει καλύτερα να ακούσετε αυτά που θα μας πει ο Σιμ Κάλλας παρά η μελέτη την οποία παρουσιάσαμε. Είχες δίκιο Μάικλ πάντως σε αυτό που είπες ότι στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και αυστηροί με τους εμπειρογνώμονες που μας παρουσιάζουν διάφορες μελέτες εδώ. Το επόμενο λοιπόν θέμα, καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο Σιμ Κάλλας. Έχουμε καθυστερήσει και εμείς, μόνο πέντε λεπτά, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, μέχρι τις 12.30 έχουμε. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πολλά εκλεκτά μέλη άκουσαν τις εξηγήσει τις οποίες θα δώσω την παρουσίαση που θα κάνω επανειλημμένα, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μειώνει ίσως τη σημασία που έχουν τα θέματα αυτά και χαίρομαι που σας παρουσιάζω τις αναθεωρη, αναθεωρημένες γραμμές και το μέσο για την συνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Έγιναν οι πρώτες προτάσεις στις 18 Οκτωβρίου και σε σχέση με την πιλωτική φάση έκδοσης των project bonds. Αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη στιγμή της οικονομικής κρίσης. Ο σωστός τρόπος χρήσης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το Connecting Europe Facility, για το συγκεκριμένο αυτό μέσο, έχουν σαν στόχο ε, τη δημιουργία ενός συστήματος μεταφορών αποδοτικού, παραγωγικού, το οποίο να επιτρέψει τη σωστή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας και των καινοτόμων μορφών συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα και με το μέσο αυτό, ταυτόχρονα και με τα ten και ταυτόχρονα και με τους στόχους για τη στρατηγική του 2020. Και αυτό καλύπτει φυσικά και την ακτοπλοεία, καλύπτει επίσης και την εσωτερική ναυσιπλοεία. Όλα αυτά θα βοηθήσουν την αποδελεσματικότητα της λειτουργίας των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 31 δις θα έλεγα είναι μια εγγύηση ότι η χρηματοδότηση θα οδηγηθεί στη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών εκεί όπου απαιτείται υψηλή προστιθέμενη αξία για τη διασφάλιση της ανάπτυξης το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe Facility δηλαδή, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να μην ζητούν από τη μία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την χρηματοδότηση των βασικών τους προγραμμάτων στα εδάφη τους και από την άλλη να μειώνουν τα ίδια τα κράτη τον προϋπολογισμό για τις επενδύσεις στα πλαίσια των πολιετών προγραμμάτων. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα κατάλογο προγραμμάτων για χρηματοδότηση στο παράρτημα στο Connecting Europe, στο μέσο Connecting Europe. Καλωσορίζω και τη δική σας πρόθεση να συνεργαστείτε με την αρμόδια επιτροπή της, με την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίσετε κι εσείς μια ισχυρή θέση διαπραγματευτική το Συμβούλιο έχει ξεκινήσει επεξεργασία των κατευθυντήριων γραμμών για τα ten Η Πολωνική Προεδρία έχει οδηγήσει σε σημαντικές συζητήσεις και η Υπουργοί στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου Μεταφορών στις 12 Δεκεμβρίου έδειξε ότι και η επερχόμενη Προεδρία της Δανίας θέλει να καταλήξουμε στα ten των οι διαπραγματεύσεις θα είναι σχετικά δύσκολες για τα μείζωνα θέματα που χαρακτηρίζουν τα ten και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των προγραμμάτων αυτών. Υψηλή προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή, διαλειτουργικότητα, αποδοτικότητα και σωστά μέσα εποπτείας. Παράλληλα, νομίζω ότι συμμεριζόμεθα την ανησυχία ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό και τα προγράμματα μπορεί να οδηγήσει σε μια πολυδιάσπαση της ευρωπαϊκής στήριξης, κάτι το οποίο θα υπονομεύσει τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε στον τομέα της, ε, των μεταφορών. Το Connecting Europe Facilities λοιπόν έχει ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Τα TEN-T's βλέπουν μέχρι το 2030 και επίσης μέχρι το 2050 για τα πολύ μεγάλα ολοκληρωμένα προγράμματα. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή ε, μεθοδολογία για τον, για τον πυρήνα της προσπάθειας. Έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση και στο εσωτερικό των κρατών μελών και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα. Καινοτομία η οποία θα περιλαμβάνει βέβαια και ε, τις υπάρχουσες υποδομές, αλλά από την άλλη θα επιλέγονται και οι προτάσεις για νέες υποδομές με υψηλή ευρωπαϊκή αξία. Θα προσπαθούμε να καλύπτουμε τους τομείς οι οποίοι ελείπουν σε αυτή τη φάση έτσι ώστε να συμπληρώνουμε τα δίκτυα και να περάσουμε από ένα patchwork πραγματικά σε ένα πραγματικό δίκτυο. Επιτροπή προτείνει επίσης ε, μια ενισχυμένη αντίληψη για τους λεγόμενους ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Αν όλα αυτά γίνονται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, τότε τα ευρώ που θα δαπανώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αξίζουν περισσότερο από το σύνολο των ευρώ τα οποία θα δαπανηθούν σε εθνικό επίπεδο. Οι νέοι αυτοί διάδρομοι, τα νέα αυτά δίκτυα θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, πολλαπλές χρήσεις μεταφορών και ε, σωστά χρονοδιαγράμματα. Είμαστε ε, αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα use it or lose it. Οι διάδρομοι αυτοί θα συνδέονται σε μεγάλες πλατφόρμες που θα αφορούν και κρατημέλη και ιδιωτικούς τομείς υπό την αιγίδα ενός συντονιστή ο οποίος θα έχει πείρα σωρεύσει από το παρελθόν. Οι πλατφόρμες αυτές στην ουσία θα ενισχύουν κάποια υπάρχοντα ήδη σήμερα φόρουμ και δεν θα οδηγούν σε περαιτέρω δημιουργία γραφειοκρατίας. Εμείς προτείνουμε πραγματιστικές επιτόπου λύσεις ανάλογα με τα μέτρα του προβλήματος κάθε φορά και όχι μια συνολική άποψη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερες εξηγήσει βέβαια για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας αυτών των διαδρόμων. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την μεγένθηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Σαν παράδειγμα θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε κάποια κενά σε υπάρχοντα δίκτυα κάποια συστήματα όπως το ΖΕΖΑΡ και άλλα και έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά χρήματα να είναι διαθέσιμα πρώτα για προγράμματα τα οποία έχουν τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. Από τα 31,7 δις που προτείνονται για τις μεταφορές, 10 αφορούν το εσωτερικό του Ταμείου Συνοχής. Τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα για τα κράτη-μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής και όχι το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ισχύσουν οι ίδιοι οι κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των Ταμείων Συνοχής, του Ταμείου Συνοχής. Είναι μια επιπλέον εγγύηση για τα επιλέξιμα κράτη-μέλη γιατί ταυτόχρονα 24 δις στη συνοχή θα έχουν άμεση σχέση με προγράμματα για τις μεταφορές. Το μέσο Connecting Europe θα καταστήσει ικανές τις επενδύσεις για τις μεταφορές του ιδιωτικού τομέα, κάτι το απαραίτητο σε περιπτώσεις δημοσιονομικής λιτότητας. Πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο ποσό θα μπορέσει να απορροφηθεί από τα υπάρχοντα μέσα ή τα προγραμματιζόμενα συγγνώμη μέσα όπως τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα project bonds. Έχουμε έτσι και αλλιώ πετύχει κάποια πρώτα θετικά βήματα με τις εγγυήσεις τις οποίες έχουμε δώσει για τη δανειοδότηση των προγραμμάτων TEN-T, ε, ιδιαίτερα στον τομέα των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας. Νομίζουμε ότι θα μπορέσουν τα χρήματα αυτά, γύρω στα 10 δις ε, της συνοχής, να λειτουργήσουν ε, με τη μόχλευση, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας άνω των 100 δις. Στο τέλος, νομίζω ότι η εκτελεστική υπηρεσία για τα τέντη θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προϋπολογισμού αυτού μέσω διαγωνισμών τους οποίους θα εκδηλώσει, θα ξεκινήσει. Αλλιώς δεν θα υπάρχει βέβαια χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάντως εσάς και την Επιτροπή σας για τη συμμετοχή σας στις 29 και 30 Νοεμβρίου στη συνάντηση στην Αμβέρσα. Αυτές οι μερίδες της Αμβέρσας επιβεβαίωσαν ότι ένας τομέας εξυγχρονισμένος με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα λειτουργήσει πίστικα για την βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές στα πλαίσια του πολιετούς οικονομικού σχεδιασμού. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ανακοίνωσε στην Ολομέλεια του μηνός Νοεμβρίου το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012-2014. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν σαν στόχο την κινητοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Να σας πω τώρα τι ακριβώς προτείνουμε για τις μεταφορές. Καθαρές μορφές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Θα κάνουμε τις πρώτες προτάσεις μας αμέσως μετά την Άνοιξη για τα καύσιμα στις μεταφορές και θα προτείνουμε επίσης και ένα νέο σιωδρομικό πακέτο μέχρι το τέλος του 2012. Θα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα και το θέμα της εσωτερικής αγοράς, τις θεσμικές μορφές διαχωρισμού ανάμεσα στους κατόχους των δικτύων και σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις γραμμές, όπως επίσης και του σιωδρομικού υλικού, του τροχαίου σιωδρομικού υλικού. Όλα αυτά με την ολοκλήρωση βέβαια των αλλαγών στον τομέα της νομοθεσίας. Και τέλος, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι θα παρακολουθήσουμε στενά τις εφαρμογές του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και τις περιοχές που έχουν κατατμηθεί. Αν δούμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, θα κάνουμε κάποιες νέες προτάσεις, πιθανώς και νομοθετικές, για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις αυτές. Ευχαριστώ, τον κύριο Επιτροπό. Εννέα αγορητές έχω στον καταλογό μου, αλλά λιγότερο από 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Δέκα οι ομιλητές. Λιγότερο από 30 λεπτά βάλε. Δύο λεπτά λοιπόν δίνω στον κάθε αγορετή και θα σας παίρνω το μικρόφωνο αν ξεπερνάτε το όριό σας. Ο κύριος Γκρός πρώτα απ' όλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Ήδη στο παρελθόν είχαμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα TNT, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και τις υποδομές για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Οπότε, επ' αυτών συμφωνούμε απόλυτα με τις προθέσεις σας και με την κρίση σας ε, για τις επιλογές που κάνετε και για τις δύο προτάσεις συμφωνούμε. Απλά να θέσω το εξής. Για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, χρειαζόμαστε κατάλληλους εταίρους. Έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή την σχετική απόφαση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση. Ε, είναι η απόφαση που πρέπει να λάβει η Επιτροπή και ουσιαστικά εξαρτάται από εσά και τον Επιτρόπο Και αφορά τα μέσα που θα πρέπει, τα κονδύλια μάλλον πρέπει να δοθούν από το Ταμείο Συνοχής. Ο δεύτερος εταίρος είναι το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι μέσα στα πλαίσια οικονομικής κρίσης αλλάζει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, οπότε πρέπει να δούμε για αυτή την πρόταση ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου. Ξέρω ότι και τις δύο προτάσεις ε, γίνονται παράλληλες συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και περιμένουμε να ακούσουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ, επαναλαμβάνω με τις προτεραιότητες που θέσατε. Και να πω ότι το 2012 θα έχουμε την ευκαιρία πλέον να συζητήσουμε και τις άλλες προτάσεις ο ενίο ευρωπαϊκός ουρανός, ναι, είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας, διότι υπάρχει η καταλεκτική ε, προθεσμή που μας πιέζει το 2012. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τελευταία στιγμή για να κάνουμε τελόγια πράξη. Θα πρέπει να δούμε γρήγορα κάποιες εξελίξεις από το κράτος μελών. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και θα με τον συνεισηγητή. Και στο δεύτερο γύρο θα καθέσω ένα ερώτημα. Well, Ayala, Η κυρία Ιάλα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κάλλας επί της αρχής στηρίζει η Επιτροπή μας, όπως στηρίξαμε και την ε, Λευκή Βίβλο για την πρόταση αυτή. Και ο νέος κανονισμός, η νέα πρόταση για τα ομόλογα έργων είναι κάτι πολύ θετικό. Βεβαίως υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη θέση των κρατών μελών που ναι μεν στις διμερείς σας επαφές σας είπαν ναι για τη λογική των ε, διαδρόμων, αλλά φαίνεται να υπάρχουν τώρα δισταγμοί και επιφυλάξεις. Θα ήθελα να ακούσω από εσά αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε με τα κράτη-μέλη, ποια είναι η στρατηγική τους και ποια είναι τα επιχειρήματα. Για το Connecting Europe, ...22 δις που είναι το ιστορικό κομμάτι των ε, δικτύων και ρωτώ όμως μετά την περαιτέρω όξυνση της κρίσης φέτος και τις περικοπές που συμφώνησε το Συμβούλιο. Ρωτώ, εν προκειμένου ποια προσθέτει η αξία για τα 10 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Συνοχής και είπατε συν 24 δις πάλι από το Ταμείο Συνοχής. Ρωτώ πώς αυτά τα επιπρόστα 10 δις που εντάσσουν στρατηγική Connecting Europe, επιπρόσθετα από τα 22 δισεκατομμύρια, πώς θα μπορέσετε να αποσπάσετε, τι αντάλλαγμα θα πρέπει να δώσετε. Έπειτα, για την ενέργεια της ελεπικοινωνίας, που είναι οι άλλοι δύο τομείς ενδιαφέροντος, πώς θα υπάρχει η κατάλληλη διάδραση. Πώς θα συνδεθούν δηλαδή οι άλλες δύο προτεραιότητες με το Connecting Europe. Ευχαριστώ, κύριε Μαϊστέρ. Τέσσερα σημεία. Καταρχάς είχαμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία μας είπε ότι σε αυτά τα ομόλογα έργων μπορούμε να πάρουμε 20, 20 περισσότερο το 20 πλάσιο από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δεύτερον, τα 230 εκατομμύρια πότε αρχίζουν ε, σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, πότε αρχίζουν μέχρι το 2013. Τρίτον, ε, είναι πολύ ευχάριστο το ότι το Συμβούλιο συζητάει τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές για τα TENS και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να συγκλίνει περισσότερο με τη δική μας θέση που είναι ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εν συνεχεία, ο διαχωρισμός μεταξύ του διαχωρισμού α, της διάσπασης των σιδηροδρόμων και του διαχωρισμού μεταξύ σειρμών και άλλων υπηρεσιών, το unbundling, ε, πότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα αυτής της αποδέσμευσης. Και τέταρτον, πρέπει όλοι να δουλέψουμε τα Χριστούγεννα και στις γιορτές και να ε, πιέσουμε τις κυβερνήσεις να μην μπλοκάρουν τους ευρωπαϊκούς ε, ουρανούς. Ο κύριος Ζέλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Σήμερα η Επιτροπή Μεταφορών πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διευκόλυνση Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, η πρόσβαση και όλα αυτά τα δίκτυα, όλη αυτή η διευκόλυνση της πρόσβασης, ότι είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε και ότι δεν θα αποκλίνουμε από αυτούς τους στόχους μας. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο θέλει να αντικαταστήσει τους διαδρόμους, το corridors, με projects, έργα. Και εμείς ε, δεν το θέλουμε, διότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πραγματικές δουλειές, πραγματικές θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Και αν μπορούμε να πάρουμε 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής, θα δώσουμε μία ευκαιρία τα κράτη-μέλη που είναι επιλέξιμα να τα χρησιμοποιήσουν και να κάνουν αυτά τα έργα. Διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε. Πρέπει να προσδώσουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυτή την αξία να την πάρουμε σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος Κράμερ, δύο λεπτά. Πρέπει εκτός όλων αυτών των καλών ιδεών να δούμε τι δεν κάναμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τώρα έχουμε περισσότερα έργα, περισσότερες αιτήσει και λιγότερα χρήματα. Θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, το αμφισβητώ. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει παράπονα και ιδίως η Γερμανία, η οποία λέει ότι χωρίς τη βοήθεια της κεντρικής κυβέρνησης, της γερμανικής κυβέρνησης, πολλά έργα δεν θα είχαν γίνει. Εγώ ξέρω παραδείγματο χάρη ότι μερικά προγράμματα όπω τα ΦΙΝ τα προγράμματα ΦΙΝ έχουν γίνει χωρίς τη βοήθεια ή χωρίς τη διαβούλευση με τους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Και στο ΕΑΤΕΜ έχετε επίσης κάτι να μας πείτε ποια είναι η βάση της σύμβασης η οποία συμφωνήθηκε και έχει υπογραφεί χωρίς τη συμμετοχή της Γερμανίας. Δεύτερον, τα μεγάλα έργα έχετε διαγράψει μερικά, αλλά ο περιβαλλοντικός τομέας είναι άμεσα συνδεδημένος με τις μεταφορές. Εάν δεν λάβουμε υπόψη την αλλαγή του κλίματος, δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Επίσης, στο, στο Δούναβι, όπου υπάρχει μεγάλη ε, ναυσιπλοεία, ε, τι θα γίνει με τη σύνδεση μεταξύ Βερολίνου και Στετίνου, δηλαδή αύξηση της ε, ναυσιπλοείας ε, στα μεγάλα ποτάμια. Λίγα λεφτά χρειάζονται και δεν καταλαβαίνω ποιος αποφασίζει πώς θα γίνει η διαχείριση αυτής του είδους της επικοινωνίας, μεταφορικής επικοινωνίας. Λίγα... Ο κύριος Κράμερ έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στη διαλειτουργικότητα. Συνδεδεμένες μεταφορές για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όμως πρέπει να προετοιμαστούμε για την... Ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων. Ποια μέτρα θα εφαρμόσει η Κομισιόν για να βοηθήσει τη διαλειτουργικότητα. Δεύτερον, αναφέρεται ότι ορισμένες χώρες έχουν αμφιβολίες όσον αφορά το δίκτυο των, ε, των διαδρόμων. Ποιε χώρε είναι αυτέ που αμφισβητούν παρακαλώ τη χρησιμοποιότητα των διαδρόμων, μπορείτε να μα το πείτε, για να μπορέσουμε και εμεί να διαφορμόσουμε την άποψή μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αναφέρεται, κύριε Επίτροπε, ότι η συμμετοχή πολλών εταίρων για τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πλατφόρμα για το θέμα των διαδρόμων που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετική αντιμετώπιση. Όμως, πιο συγκεκριμένα, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα στελεχωθεί, πώς θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα των διαδρόμων. Δεύτερον, έχετε μια στρατηγική να αντιμετωπίσετε τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αμφιβολίες και αμφισβητούν τη χρησιμότητα αυτής της πρότασης. Και αν έχετε στρατηγική, ποια είναι, παρακαλώ, πέστε μας. Και τρίτον, πώς θέλετε να διαμορφωθεί συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν των αρμοδίων συντονιστών και της πλατφόρμας των διαδρόμων, αυτού του δικτύου διαδρόμων. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάβεσαρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διαθέσή μου, οπότε δεν μπορώ να τεκμηρώσω πλήρως το ερώτημα που θα θέσω. Ήδη εξέφρασαν οι συνάδελφοι τη θέση του σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και με το Connecting Europe. Η θέση των κρατών μελών ε, ήταν σαφή στο τελευταίο Συμβούλιο Μεταφορών. Πάντω, θα θέσω ένα ερώτημα που ήδη έχει ξανακουστεί. Σχεδιάζετε να κάνετε κάτι στους κόλπους Επιτροπής ε, για να ανατρέψετε την θέση ε, στο Συμβούλιο ε, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Χαιρετίζω τα σχόλια του Επιτρόπου για το ΣΕΖΑΡ. Με ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να συνεργαστεί στενά με τον Επίτροπο για να επιτύχουμε πρόοδο στον ε, ευρωπαϊκό ουρανό. Επίση, για τη χρηματοδοτική στήριξη του project είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ορθά είπατε, πρέπει να δούμε την προσθέμενη του αξία. Όλοι να γνωρίζουμε ότι σε όλη την Ένωση, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ε, συμφόρησης, ε, ιδίως ερωλημένε. Εγώ θα είμαι εισηγήτρια ε, για αυτό το φάκελο και, όπως είπα και πριν, το μήνυμα που θα προσπαθήσει να περάσει με την επόμενη χρονιά η Επιτροπή μας είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος... Ε, μάλλον οι συνάδελφοι έθεσαν πολύ εύστοχα ερωτήματα, οπότε να μην θέσω εγώ ερώτημα. Καλύτερα να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Κυρία Στεναλόβα. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για την διάθεσή σας να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση ε, στην Επιτροπή μας. Και πιστεύω ότι και η συζήτηση με κρουσόπους των μελών είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπατε, use it or lose it. Θεωρώ και εγώ ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχή και πρέπει να δούμε πώς λειτουργήσει πρακτικά. Λέω, αν αποτύχει αυτό το project, δεν θα μπορεί κανείς να τλήσει τα κονδύλια από τα Ταμείο συνοχή, Ρωτώ, συγκεκριμένα, έπειτα, οι κανόνες είναι απόλυτα σαφή σχετικά με τους τρόπους που θα γίνεται η συγχρηματοδότηση. Έπειτα, πώς θα γίνεται η επιλογή των project με υψηλή προστιθεμένη αξία, ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσει. Πώς θα καθορίζεται αυτή η ε, υψηλή προσταμένη αξία. Και θα προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Επίσης έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας βαθμός δυσπιστίας εναντί των νέων κρατών μελών. Ελπίζω ότι με τον νέο μηχανισμό ενισχυθεί η αμοιβή εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ η κυρία Σαρακιάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο επίσης. Δράτω με της ευκαιρίας για να επενθυμίσω μόνο το εξής. Το 2012 θα είναι ένα έτος κατά το οποίο θα μας απασχολεί και η διαπραγμάτευση για την αδιατύπωση της πρότασης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει μια αποτελεσματική ε, στάση στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο και καλούμε τον Επίτροπο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ειδικό πολιτικό του βάρος ώστε να πείσει τις εθνικές κυβερνήσεις ότι θα πρέπει το πρώτο εθνικό πακέτο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να ληφθούν και μέτρα ε, σε περίπτωση που συμβεί το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών σαν να κάναμε τον, τα 100 μέτρα sprint. Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να μείνετε στο χρόνο που σας έδωσα, οπότε θα δώσουμε 10 ε, λεπτά στον Επίτροπο να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που ετέθησαν. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, <coughs> σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις για κάποια θέματα που φαίνεται να αφορούν πολύ κόσμο. Κύριε Κράμερ, είπατε ότι κάποιοι παραπονούνται ότι τα προγράμματα επελέγησαν χωρίς τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είχαμε δύο ολόκληρους γύρους διαπραγματεύσεων με όλες τις κυβερνήσεις. Από την αρχή είχα φοβηθεί ακριβώς ότι θα αρχίσουν να μας πιέζουν για να προωθήσουμε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα εις βάρος άλλων. Και πράγματι άρχισαν να θέτουν θέματα όπως αυτό γιατί δεν το επιλέγετε, αυτό γιατί δεν το επιλέγετε κτλ. Όταν κάποιος έρχεται και παραπονείται, ε, εγώ ε, δεν δέχομαι ότι αυτό σώνει και καλά είναι κάτι το πάρα πολύ καθοριστικό και αφορά κάτι το οποίο κάναμε και δεν το κάναμε καλά. Πάντως υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα τα οποία έχουν επανειλημμένα τεθεί και στο Κοινοβούλιο και σε άλλα ε, όργανα όταν συζητάμε τα θέματα αυτά. Σαν παράδειγμα όταν συζητήσαμε το θέμα του αρκτικού λεγόμενου διαδρόμου. Λοιπόν, δύο θέματα. Από τη μία η διάδρομη, από την άλλη τα δεκαδείς. Το θέμα είναι τι θα γίνει σαν παράδειγμα αν δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που είναι διαθέσιμα. Απλά θα εφαρμοστούν οι κανόνες. Γιατί τους κανόνες τους ελέγχει ακόμα και η Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και μπορεί εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για την εκ νέου χρήση τους. Αυτά έχουν συμβεί και σε σχέση με τα τεντής. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία νομοθετική η οποία είχε προταθεί στις 19 Οκτωβρίου με τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν είμαστε ακόμα απόλυτα έτοιμοι Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Connecting Europe Facility, στο μέσο Connecting Europe, αλλά η διαδικασία ιδιαίτερα των project bonds δεν έχει όπως ξέρετε ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τα μέσα για να μπορέσουμε να περάσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν γενικότερα θέματα, διάδρομοι, πώς τους διαχειριζόμαστε τους διαδρόμους. Το θέμα της διαχείρισης ή ε, διακυβέρνησης εισαγωγικά των ε, διαδρομών περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές σε αρκετό επίπεδο λεπτομέρειας. Είμαστε ευέλικτοι όταν συζητάμε τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία αυτών των διαδρόμων. Θέλουμε βασικά να αποτρέψουμε γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και επικαλύψεις ακούμε τα σχόλια και τις προτάσεις, προσπαθούμε κάποιες από τις προτάσεις αυτές να τις χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιούμε και τις εθνικές ή κυβερνητικές δομές όπου αυτές προσφέρονται, αλλά οι διάδρομοι κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε ένα πρόωρο αν θέλετε, σε ένα πρόωρο στάδιο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις θα ανατρέψουμε ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. οι διάδρομοι όταν τους βλέπει κανείς στο χάρτη αυτή είναι η ουσία αν θέλετε της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Βλέπετε ότι αυτές οι ροές οι μεταφορικές έχουν οικονομική σημασία, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και εδώ βρίσκεται η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Αλλά όπως είπα είμαστε ευέλικτοι Το αν θα συζητήσουμε λεπτομέρειες σαν παράδειγμα το στετίνο θα συμπεριληφθεί στο διάδρομο ή θα εξαιρεθεί του διαδρόμου. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, διακλαδώσεις χωρίς όμως να χάσουμε τη βασική μας γραμμή, την βασική εικόνα. δεν θέλουμε να υπάρχει σύγχυση επίσης ανάμεσα ε, στους διαδρόμους και σε επιμέρους μικρότερα δίκτυα. Αυτό θα ήταν μια αποτυχία. Ακολουθούμε λοιπόν μια συγκεκριμένη στρατηγική για να υπερασπιστούμε τη λογική των διαδρόμων. Πάντως, αν κάποια άλλη πλευρά κάνει προτάσεις, σεβόμενες προτάσεις στις κοινέ αξίες τις οποίες έχουμε, σε αυτή την περίπτωση θα εξετάσουμε τις προτάσεις να το γνωρίζετε αυτό, δεν αγνοούμε καμία πρόταση αλλά θα πρέπει να εντάσσεται η πρόταση αυτή στην ευρεία εικόνα αν θέλετε γιατί δακτύλοι λείπουν δεξιά και αριστερά στους διαδρόμους. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Υπάρχουν επίσης ε, και πάρα πολλά προβλήματα συνοστισμού ε, μεταφορικών δικτύων και ροών. Δεν μπορούμε μέσα από τους διαδρόμους να τα λύσουμε όλα αυτά. και θυμίζω ότι χρησιμοποιούμε κυρίως τις εθνικές υπάρχουσες δομές. Λοιπόν, για τα δέκα δις. Τα 10 δις λοιπόν. Εδώ θα εμείνω θα έλεγα, θα είμαι πισματάρης και θα υπερασπιστώ τις προτάσεις αυτές τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι τελευταία γρανίδος. Όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και σε επίπεδο συμβουλευτικών επιτροπών και σε επίπεδο συμβουλίου ενισχύουν την άποψη που έχω ότι πρόκειται για το σωστό μέσο. Αν θέλετε στις παρατηρήσεις που έκανα σήμερα, δεν ξεκαθάρισα ίσως απόλυτα ότι τα χρήματα αυτά έχουν φύγει ε, από, δεν είπα ότι έχουν φύγει τα χρήματα αυτά από το συνοχή. Δεν, το αντίθετο συμβαίνει. Τα τέντη είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη. Οπότε μιλάμε για ένα ποσό το οποίο έχει σαν στόχο ένα συγκεκριμένο μέσο για μια συγκεκριμένη κατηγορία χωρών, τις χώρες συνοχής. Χθε συνάντησα πολλούς δημοσιογράφους και τους είπα ότι αυτό το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ είναι το εξής. Αν πιστεύετε ότι αυτές οι προτάσεις δεν είναι αποδεκτές και αν υπάρχουν διαφωνίες από πλευράς των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ξέρετε ότι θα έχουμε προβλήματα και συζητήσεις έντονες, σαν παράδειγμα με την Περιφερειακή σας Επιτροπή. Τότε θα πρέπει να αναπέμψουμε το θέμα στο Συμβούλιο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο θα πάρει τα χρήματα και δεν ξέρω τι θα τα κάνει, μπορεί και να τα εξαφανίσει, να τα σκορπίσει. Ας πούμε ότι δεν δέχεστε σαν παράδειγμα για το μέσο Connecting Europe να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά από τα 10 δις. Δικαίωμά σας, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά από την άλλη, αυτό που δεν θέλω να δω να συμβαίνει είναι αυτά τα 10 δις τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό του Connecting Europe να πολυδιασπώνται με εθνικά, τοπικά, περιφερειακά συμφέροντα, να διαλύονται όλα αυτά. Να υπάρχει μια τέτοια διασπορά που να εξαφανίζονται τα χρήματα αυτά και να ενσωματώνονται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο σε εθνικούς προϋπολογισμούς μέσω της κονιορτοποίησής τους. Αυτό δεν θα ήθελα να συμβεί. Αρκετά μέλη ρώτησαν γιατί αυτή η επιλογή για τα 10 δις ε, ξεχωριστά. Εγώ νομίζω ότι ακριβώς στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης, η κοινή διαχείριση ξέρετε είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και εξυπηρετεί και κάποιες εθνικές προτεραιότητες και το Ταμείο Συνοχής στις εθνικές προτεραιότητες έχει παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά εδώ μιλάμε για προστιθέμενη αξία προστιθέμενη αξία η οποία θα εξυπηρετήσει ακριβώς τις διασυνδέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά σημεία της Ένωσης. Η στρατηγική για την υπεράσπιση λοιπόν αυτός, αυτής της λογικής ε, θα προέλθει από εμά. Υπάρχει σκληρή κριτική από τις λεγόμενες χώρες Βίσεγκραντ. Οι εκπρόσωποι των χωρών Βίσεγκραντ, ιδιαίτερα από την τσεχική κυβέρνηση, έχουμε διαφωνίες Έχουμε συμφωνήσει στο ότι στις αρχές του επομένου έτους θα έχουμε μια συνάντηση μαζί τους και θα προσπαθήσουμε να τους παρουσιάσουμε την ιδέα αυτή με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο, προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε για το πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά, πώς μπορούν οι ίδιοι να κάνουν προτάσεις για χρηματοδοτήσεις, θα σταθούμε ελαστικοί, ευέλικτοι Και ξέρετε ότι μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι το 85% το επίπεδο χρηματοδότησης. Αλλά όταν λέω μέχρι το 85% το εννοώ, δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι στο 85%. Μέχρι το 85%. Υπάρχει λοιπόν μία πρόταση σε σχέση με το 2,5 του ΑΕΠ για να υπάρξει διαφορετική στήριξη και πάντα εμείς θεωρούσαμε ότι αυτά τα, τα 10 δις είναι εκτός αυτής της προϋπόθεσης. Δεν μπορεί να έχετε τρεις χώρες για ένα πρόγραμμα και μία χώρα να έχει απορροφήσει το 2,5% και να μην μπορεί να συνεχίσει, ενώ οι άλλες χώρες να θέλουν να προχωρήσουν. Όλα αυτά είναι περισσότερο οικονομοτεχνικά βέβαια και γι' αυτό θα τα κατανοήσετε όταν τα δείτε γραμμένα στα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει θα διευκρινιστούν όλα αυτά. Το βασικό θέμα για σας και για τα κράτη-μέλη βέβαια σε αυτή τη φάση είναι ο συνδυασμός της επικουρικότητας από τη μία με, την, με τον κοινοτικό χαρακτήρα από την άλλη. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα μπροστά μας το οποίο να είναι δεσμευτικά δεκτό από τα κράτη-μέλη. Εφόσον υπογράψουν θα πούνε ναι τελείωσε, θα γίνει αυτός ο διάδρομος και εφόσον υπογράψουμε θα εφαρμόσουμε και θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Όλα αυτά χρειάζεται να διευκρινιστούν σε επίπεδο λεπτομέρειας και μέσω της νομοθετικής προσπάθειας που θα ακολουθήσει για να καταλήξουμε στις βέλτιστες δυνατές λύσεις, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε για τη συνεισφορά του γενικότερα και για τη συντομία. Μπορέσαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σε περισσότερες ερωτήσεις. Έχουμε θέματα φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πείσουμε την Περιφερειακή Επιτροπή ότι δεν είμαστε ληστές και θέλουμε να κλέψουμε τα χρήματά τους, αλλά θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μεταφορών. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Πριν εξαφανιστείτε όλοι, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσά και στο προσωπικό σα καλά Χριστούγεννα κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στα μέλη ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε μία ακρόαση, ακρόαση γιατί για τους ταχογράφους. Εκτιμώ ότι τα μέλη έχουν άλλα σημαντικά πράγματα να κάνουν, αλλά δεν θέλω να είμαι εδώ με την κυρία Τίκα, εγώ και 100 εμπειρογνώμονες και όλα τα έδρανα των ευρωβουλευτών να είναι άδεια και να έχουμε μόνο τους εμπειρογνώμονες, τους ακροατές και έχουμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα των ταχογράφων και μετά τα πλοία διπλού κήτου στο τέλος. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα καυτά θέματα. Ξέρω ότι θα έρθείτε όλοι εδώ και θα κάνετε το χρέος σας.